Colleagues, first of all, Happy ε, καταρχήν καλή χρονιά για όσους δεν σας ευχήθηκα ακόμα. Στο καλή χρονιά εύχομαι και στο, προσωπικό του Ευρωκοινοβουλίου και στους διερμηνείς και σας ζητώ καταρχήν να κοιτάξουμε και να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσης διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά έχουμε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 26 25-26 ε, Νοεμβρίου και πάμε στη σημερινή μας ημερήσια διάταξη που έχουμε το ε, πρόγραμμα Ναϊάδες 2, ε, το πρόγραμμα δηλαδή για τη στήριξη των πλωτών οδών και την μήνυα κρόαση Εξήγησα μόλις του συνάδελφου εδώ στο έδρανο ότι οι βουλευτές είναι πάντοτε ενθουσιώδεις για τις ακροάσεις, γιατί πρέπει να κάνουμε ακροάσεις και να φέρνουμε τους ε, ειδικού, ε, αλλά στην πράξη πολύ λίγοι ε, εμφανίζονται στις συνεδριάσεις. Είναι μια από τις αδυναμίες της λειτουργίας εδώ του σώματος. Ελπίζω πως και άλλοι θα έρθουν αργότερα. Η κυρία Βόρτμαν Κόλτ, η συγκίτρια που ε, μας ζητά συγγνώμη που είναι απούσα, η, το, το, το, η ακρόαση αποτελείται από δύο πάνελ. Το ένα αφορά τη βέλτιστη ε, ολοκλήρωση των, των εσωτερικών πλωτών οδών, ε, στο σύστημα μεταφορών και ένα δεύτερο πάνελ με τις εσωτερικές πλωτούς, πλωτές οδούς και πάλι με τέσσερις εμπειρογνώμους. Ο κάθε εμπειρογνώμονας έχει 6 λεπτά για την εισηγήσή του και μετά θα έχουμε ερωταπαντήσεις. Χωρίς άλλη καθυστέρηση. Θα περάσουμε στο πρώτο τμήμα που τιτλοφορείται... Α, συγγνώμη, καταρχήν έχουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλο ξεχνάω. Αλλά δεν πειράζει, μας θυμίζουν εκείνοι. Έχουμε λοιπόν εκπρόσωπο της DG Move. Κομισιόν. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο που διοργάνωσε αυτή την ακρόαση υπέρ της ανάπτυξης της, εσωτερική, της πλοήγησης εσωτερικών υδάτων. Ε, και με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τις εισηγήσεις των πυρογνωμόνων. Ε, σύντομα θα σας παρουσιάσω αυτό το πρόγραμμα Αναγιάδες 2, είναι το δεύτερο τέτοιο πρόγραμμα το περασμένο συμπεριλάμβανε διάφορες δράσεις σε πέντε τομείς με διάφορες δράσεις ο καθένας και τώρα είναι ο διάδοχος του πρώτου προγράμματος όπου το βασικό που θέλαμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε τις προσπάθειες όλων σε έναν περιορισμένο ρυθμό δράσεων. Το πρόγραμμα ΝΑΕΔΕΣ 2 είναι προσανατολισμένο στη δράση και παρακαλώ να μην κρίνετε το πρόγραμμα από τις δύο νομοθετικές προτάσεις που έχετε ενώπιόν σας, γιατί είναι μόνο η αρχή. Ε, το ένα είναι η πρόταση για την καλύτερη χρήση του αποθεματικού, όπως αποκαλείται, δηλαδή διορθωτικά μέτρα. Και το άλλο είναι ε, οι προπαρασκευαστικές δράσεις για να εισαχθεί το νέο σχέδιο ε, διακυβέρνηση που προτείνουμε. Όμως υπάρχουν πολλά μέτρα ε, που προετοιμάζονται σε σχέση με το θέμα της ποιότητας Έχουμε λοιπόν υποδομές, καινοτομία, αγορά, περιβάλλον, ε, ε, θέσεις επασχόλησης, δεξιότητες και πολυτροπική ολοκλήρωση. Ε, έχουμε διάφορες δράσεις που βλέπετε για κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες. Τώρα όσον αφορά το θέμα των υποδομών, που βεβαίως είναι ε, το βασικό προαπαιτούμενο για να μπορεί να λειτουργεί ένας τρόπος μεταφορών, αυτό που προτείνουμε είναι η εξαιρετική ε, ολοκλήρωση των ε, εσωτερικών πλωτών οδών στο νέο πολυ ε, το, ε, το, το, νέο πρόγραμμα με πολλά εκατομμύρια ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το Horizon 2020. Έτσι θα υπάρξουν νέα, νέοι πόροι προς όφελος αυτού του τομέα και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες ξεπερνούν αυτό που λογικά θα ανέμενε κανείς από ένα στάνταρ πρόγραμμα. Οπότε θέλουμε και προτιθέμεθα να κερδίσουμε εκμεταλλευόμενοι όλα τα μέσα χρηματοδότησης που δίνουν διαθέσιμα για τις ναϊάδες, αντί να έχουμε μια περιορισμένη οροφή. Όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς και την περιβαλλοντική ποιότητα της ε, πλοήγησης ιστορικών οδών, αυτό θα ωφελήσει ε, και για τις υπηρεσίες της αγοράς αυτής ε, που και έχουμε επαφές με τους εκπροσώπους του φορέα, του τομέα μάλλον, ε, για να μας πούν ακριβώς τι χρειάζονται για να στοχεύσουμε και εμείς μέσα ε, στήριξης για τις βιώσιμες υπηρεσίες μεταφορών στους νέους διαδρόμους μεταφορών. Ε, επίσης ε, σκοπεύουμε να κάνουμε μια γενική μεταρρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας. Θα είναι σίγουρα κάτι το σημαντικό για την επόμενη Κομισιόν, εσωτερικές πλωτεσόδη, δεξιότητες, αλλά και κοινωνικές πτυχές όπως αυτές που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά και τα πληρώματα. όχι μόνο για τους ε, καπετάνιους των ε, ε, καραβιών αλλά για ολόκληρα τα πληρώματα. Δεύτερο θέμα είναι το, η βελτίωση των υπηρεσιών ε, ενημέρωσης ε, για τους ποταμούς έτσι ώστε αυτές οι υπηρεσίες να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και να ενταχθούν πλήρως στις μεταφορές. δεν μπορούμε να πάμε από την πόρτα του εργοστασίου στην πόρτα του καταναλωτή εάν δεν χρησιμοποιηθούν συνδυασμένα οι μεταφορές και οι πλωτές οδοί μέσα σε αυτές. Μετά δηλαδή από την ε, στήριξη, μάλλον μετά από την ασφάλεια και τις επιχειρήσεις, τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για, για την ε, υποδομή, την ηλεκτροτεχνική υποδομή ώστε να ολοκληρωθούν αυτές, να ενταχθούν αυτές οι πλωτές οδοί στο ολοκληρωμένο σύστημα. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται συντονισμένες δράσεις και γι' αυτό και έχουμε προβεί σε ένα μέγα άνοιγμα προς τις επιτροπές των ποταμών River Commissions. Μόνο αν μπορέσουμε να ε, ε, τυθασεύσουμε όλες τις εξουσίες όλων των οργανισμών που εργάζονται για τις εσωτερικές πλωτές οδούς θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα απτά. Και θα ήθελα να στείλω ένα προσωπικό χαιρετισμό στους εκπροσώπους του τομέα που είναι μαζί μας ε, σήμερα. Επίση, ο ίδιο ο, το, θα πρέπει να κάνει κάποια βήματα, να ολοκληρωθεί, να ενσωματωθεί περισσότερο. Θα ήταν ε, ουτοπικό να φανταστούμε ε, ε, μέτρα στήριξη ανά σκάφος. Αυτό δεν γίνεται. Η μόνη δυνατότητα για να μπορέσει να απελευθερωθεί η χρηματοδότηση θα είναι εάν ο ίδιο ο τομέα μπορέσει να ολοκληρωθεί και να σχηματίσει τι σωστέ δομέ, ώστε να μπορεί να λάβει και να απορροφήσει τη χρηματοδότηση. Όπως γνωρίζετε, οι δύο προτάσει. που υποβάλλουμε τώρα είναι ε, μια που είναι επίγουσα και είμαστε πολύ ευγνώμονες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ασχολείται με αυτό το θέμα όσον αφορά την απελευθέρωση του αποθεματικού που απαντά έτσι στην κρίση και το δεύτερο είναι η νέα διακυβέρνηση που θα είναι πολύ σημαντική και να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα μόνο χώρο εσωτερικής πλοήγησης στο σύνολο της Υπήρου, όχι μόνο στο Δούναβι βιτορινο αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. για να μπορέσουμε να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά, αποδοτικά. Θα, όσον αφορά τις εκθέσεις, θέλαμε να συγχαρούμε την εισηγήτρια του Κοινοβουλίου που έχει κάνει εξαίρετη δουλειά μέχρι τώρα. Έχουμε βεβαίως κάποια σχόλια που θα θέλαμε ε, να αναφερθούν ναι, πετήσεις για λιγότερη γραφειοκρατία θα πρέπει να εφαρμοστούν και για την Κομισιόν όσον δηλαδή τι αναφορέ κτλ. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες στις οποίες θα επανέλθουμε ε, εν ευθέτω χρόνο. Αν γίνει θα ήθελα να πω πως ε, ε, πρέπει να σας ευχαριστήσω όλους γιατί συμμετείχατε στη μακρά διαδικασία διαβούλευσης που οδήγησε στη δημοσίευση του προγράμματος Ναϊάδες τώρα. Ήμασταν σε επαφή ε, τα τελευταία τρία χρόνια. Πέρυσι φτιάξαμε το έγγραφο εργασία για το Ναϊάδες και τώρα βέβαια το νέο πρόγραμμα Ναϊάδες αποτελεί την υλοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής της ε, μακράς ε, και μεγάλης κλίμακας διαβούλευσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εδώ σταματώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Θεολογίτη και πάμε αμέσως στην ακρόαση στο πρώτο τμήμα ε, με τίτλο «Προς μια ολοκλήρωση των εσωτερικών πρωτονοδών». Έχουμε πέντε ομιλητές Έρικ Σταφ που είναι επικεφαλής ε, της Συμμαχίας ε, Ευρωπαϊκών Υποδομών, τον το κύριο Μάζικ που είναι Γενικός Διευθυντής ε, της Επιτροπής του Δούναβη και, και κύριο Κρότ που είναι Γενικός Γραμματέας της North International εξ του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Μεταφορές. Έχουμε λοιπόν 6 λεπτά για κάθε ε, εισηγητή. Έχετε, Κάριν, το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή χρονιά σε όλους σας. Η εσωτερική ναυσιπλοεία, η οργάνωση εσωτερική ναυσιπλοεία τη Ευρώπη είναι κυρίω δημόσιο φορέα. Είμαι δημόσιο φορέα, μάλλον απαρτίζεται και από δημόσιου φορέα και προσπαθούμε να έχουμε καλύτερη και βιώσιμη κινητικότητα και είναι πολύ σημαντική ε, πτυχή η εσωτερική ναυσιπλοεία και θεωρούμε ότι αυτή η ποταμή ε, είναι ένα εργαλείο αλλά έχει αυτός σκοπός. Λοιπόν, είναι λογικό να έχουμε πιο αποδοτική κινητικότητα των ανθρώπων, αλλά είναι εξίσου λογικό να έχουμε πιο αποδοτική κινητικότητα των φορτίων. Και θα μπορούσατε να έχετε μεταφορά ε, μέσω πλοίων, μέσω τρένων. Πρέπει να κάνουμε πολλά, να δούμε ποιο το δυναμικό που διαθέτουμε και, για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι πολλοί πλειοκτήτες ε, έρχονται σε εμά και πολλοί μεταφορείς έρχονται σε εμά και θέλουν να χρησιμοποιούν τις οδούς εσωτερικής νευσοπλοείας και θέλουν να ε, χρησιμοποιήσουν ένα τμήμα αυτής της αλυσίδας είναι νέοι χρήστες, δεν ξέρουν το σύστημα και δεν είναι οι πολύ γνωστές εταιρείε. Και αυτό είναι ένα σημάδι ότι ίσως να υπάρχουν και νέοι πελάτες, αλλά αλλάζει και η οικονομία στην Ευρώπη. Η βαριά βιομηχανία φεύγει από τους ποταμούς Μεταφορά άνθρακος μειώνεται, χάλιβα μειώνεται. Άρα βλέπουμε μεγάλη ριζική αλλαγή. Προσπαθούμε οι νέοι μεταφορείς που χρησιμοποιούν πλοία να έρθουν σε επαφή με τους προμηθευτές για να καλύπτονται οι ανάγκες τους. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Άρα πρέπει να κάνουμε αλλαγές και πρέπει να διαμορφώσουμε σωστή πολιτική συστημική πολιτική απαιτείται. Όχι μόνο με τρόπους μεταφορά συνδέεται, πρέπει να λειτουργεί η ναυσιπλοεία εσωτερική στο σύστημα βέβαια, αλλά θέλουμε να λειτουργεί η ναυσιπλοεία εντός του γενικότερου συστήματος. Αν θέλουμε να έχουμε την ε, προσέγγιση διαδρόμων που έχει σχεδιαστεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβουλίο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις πτυχές. Όπως τις υποδομές, ψηφιακές υποδομές για διαβίβαση πληροφοριών και για κοινή χρήση μεταφορικών μέσων. Λοιπόν, να αρχίσουμε να ομαδοποιούμε τα φορτία. Χρειάζεται βελτιστοποίηση των φορτίων, πολλή συνεργασία. Γίνεται πιο περίπλοκη η κατάσταση και νομικά και σε άλλους τομείς πρέπει να εξετάσουμε την νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ενεργειακή χρήση για τις μεταφορές, η ένταση της χρήσης ενεργείας να μειωθεί και το ίχνος του άνθρακα να μειωθεί. Πρέπει να δούμε και το κόστος. Το κόστος των υποδομών, το εξωτερικό κόστος. Δεν θα πρέπει να τα βάζουμε όλα σε ένα καλάθι να χρησιμοποιούμε σωστά όλα τα διαθέσιμα μέσα. Και η εσωτερική ναυσιπλοεία πρέπει να χρησιμοποιηθεί βέβαια. Έχουμε το ΝΑΙΑΔΕΣ 2 και έχουμε ένα πρόγραμμα από το 2014 το 2020. Άρα είναι σημαντικό να εφαρμοστεί. Ποιε είναι οι δικέ μα ύψε προτεραιότητε, οι σκληρέ υποδομέ, ευφυεί υποδομέ χρειαζόμαστε, βιώσιμε υπηρεσίε και καινοτόμες τεχνολογίες. Η σκληρή υποδομή είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Στο Κοινοβούλιο κάνατε θαυμάσια δουλειά. Έχουμε συμπεριλάβει τους σημαντικούς ποταμούς στους διαδρόμους με, τη με το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης μπορούμε να κάνουμε επιτέλους δουλειά. Έχουν οριμάσει πολλά προγράμματα που έχουν δρομολογηθεί και το υψηλό ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι ε, το κίνητρο για να συνεργαστούν οι κυβερνήσεις. Έχουμε και πολιτικός πώς, πιο δύσκολα προγράμματα και εκεί έχετε ρόλο να βγούμε από το τέλμα και από τη στάθμιση ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την επιμελητία της εσωτερικής ναυσιπλοείας και πώς μπορούμε τις εσωτερικές ε, υδάτινες οδούς να τις κάνουμε να τις χρησιμοποιούμε με διάφορους ποικίλου τρόπους. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και από τα πολιτικά ευαίσθητα προγράμματα να κινηθούμε προς σωστή εφαρμογή της εσωτερικής ναυσιπλοίας Το ψηφιακό τμήμα. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, το κατάλληλο. Πρέπει να εφαρμοστεί σωστά το πλαίσιο. Και να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια για, την, για το ψηφιακό προγραμματισμό. Για τις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στο ΑΤΕΝΤΗ και στο ΣΕΦ, αλλά έχουμε, έχετε μπροστά σας δύο νομοθετικές προτάσεις, έτοιμες. Δεν χρειάζονται πολλές αλλαγές. Θα ήταν πολύ καλό αν πριν τις εκλογές τα προωθήσετε αυτά τα ζητήματα. Αυτά έχω να πω για την ώρα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Κάρεν. Προχωράμε στον Έρικ Στακ. Επί κεφαλής της Συμμαχίας για την Ευρωπαϊκή Επιμελητία και Οργάνωση των Δικτύων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Σας έχω φέρει ορισμένες διαφάνειες στα αγγλικά βέβαια, αλλά εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Θα αρχίσω αναφέροντας σας ορισμένες ε, πτυχές που αφορούν ιδιαίτερα τον ε, τομέα της ε, εφοδιαστικής και της διαχείρισης της διακίνησης. Κέντρο του ενδιαφέροντός μας είναι να θεωρούμαστε ένα συστατικό στοιχείο του συστήματος της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ εύκολο, όμως είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των κάθε, του κάθε λιμάνιου και του κάθε κρατούς ε, μέλους. Τα λιμάνια λοιπόν, τα εσωτερικά λιμάνια ε, ανήκουν στο σύστημα και να σας πω ότι έχουν δημιουργηθεί νέες προοπτικές. Και αυτό καθιστά αναγκαία την καινοτομία. Η εσωτερική ναυσιπλοεία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο στον ε, τομέα των, ε, της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Όμως, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Τα εμπορευματοκιβώτια δεν ε, μπορούν εύκολα να μεταφερθούν από τους εσωτερικούς ελιμένες ε, στα ε, τρένα, στους σιδηροδρόμους. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται βελτίωση, βελτίωση που θα έρθει μόνο με την καινοτομία. Τώρα, προβλήματα και συμφόρηση παρατηρούνται στο εσωτερικό δίκτυο ναυσιπλοείας, ιδιαίτερα ανάμεσα στο Δούναβι και στον Ρήνο. ιδιαίτερα στην περιοχή, για παράδειγμα, του Στράουμπιν της ε, Βαβαρίας. Και να πω ότι χωρίς ε, την ε, βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου δεν θα μπορέσουμε να βρούμε μια κατάλληλη λύση έτσι ώστε η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων στους, στις εσωτερικές πιλωτές οδούς να γίνει πιο αποδοτική. οι μεταφορές στις εσωτερικέ απλωτές οδούς θα αναπτυχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως είπα, εάν ενσωματωθούν στο διατροπικό δίκτυο μεταφορών. Γι' αυτό το λόγο εσείς πρέπει να θεωρείτε ε, εμάς ως έναν σημαντικό εταίρο και όχι ως ανταγωνιστή. Πρέπει να υποστηριχθούν και να προωθηθούν νέες διατροπικές υποδομές που θα συνδέουν πολλούς μεταφορείς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζονται να δημιουργηθούν προϋποθέσεις υποδομής μεν, όμως αυτό θα γίνει μόνο με την δημιουργία ενός πραγματικά διατροπικού αποδοτικού δικτύου μεταφορών. Θα σας ε, παρουσιάσω τώρα το δίκτυο που έχουμε αναπτύξει στο Duisburg, όπως βλέπετε στο, στην αριστερή διαφάνεια, μέσω του οποίου συνδέουμε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Τα οι περισσότερες συνδέσεις Ευρώπης ε, και Ανατολής Κίνας, για παράδειγμα, συνδέονται από το λιμάνι του Τούσποκ, ένα εσωτερικό λιμάνι, και όχι, για παράδειγμα, από το λιμάνι του Αμβούργου, που βρίσκεται πιο κοντά στη θάλασσα. Έχει, λοιπόν, ε, ιδιαίτερη σημασία το εσωτερικό αυτό λιμάνι. Τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε δραστηριοποιηθεί και συνεργαζόμαστε με πολλές βιομηχανίες. Για παράδειγμα με την ε, αυτοκινητοβιομηχανία Audi, η οποία παράγει ορισμένα εξαρτήματα που σε εργοστάσιο κοντά στο λιμάνι μας και από εκεί αποστέλλονται σε όλο τον κόσμο, στα εργοστάσια συναρμολόγησης. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα του μεγέθους του όγκου ε, που διακινούμε, διακινούμε κάθε μέρα φεύγει ένα ολόκληρο κοντέινερ από το λιμάνι μας, γεμάτο με μηχανές, το οποίο κατευθύνεται από τη Βαβαρία σε εμάς, στο Duisburg και από εκεί σε όλους τους ε, προορισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η σωστή και γρήγορη σύνδεση σιδηροδρομικού δικτύου με ε, εσωτερικής πλώτης οδού. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι, το, είναι η στάθμη των υδάτων των ποταμών. Το 2003 που είχαν παρατηρηθεί προβλήματα με τη στάθμη του Ρήνου, είχαμε αναγκαστεί να βρούμε επίγουσες λύσεις και να μεταφορτώσουμε όχι στο που αλλά στο Λούντβιξ Χάφεν, πιο νότια. Χρειάζεται λοιπόν μία προσέγγιση με νέες ιδέες, με ένα ολόκληρο κόνσεπτ το οποίο θα είναι υλοποιήσιμο. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Κάθριν Όμπστ, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εσωτερικών Λιμένων. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να παρουσιάσω την δική μας άποψη για το πρόγραμμα ΝΑΙΑΔΕΣ. Εμείς αντιπροσωπεύουμε 200 λιμένες σε 19 χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σκεφτόμαστε το νερό όταν γίνεται λόγος για εσωτερικούς λιμένες. Είναι όμως ε, πολύ σημαντικό να δούμε και ε, τι κρύβεται πέρα από αυτό. Τις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις. οι οποίες χρειάζονται έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά του φορτίου. Η βιομηχανία επίσης εξαρτάται απόλυτα από τα δίκτυα αυτά, τα διατροπικά δίκτυα. Ορισμένα γενικά σχόλια για το πρόγραμμα ΝΑΙΑΔΕΣ. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εσωτερικών Λιμένων στηρίζει τον ε, γενικότερο στόχο του προγράμματος ε, ΝΑΙΑΔΕΣ 2, δηλαδή να βελτιώσει και να δημιουργήσει συνθήκες για την βέλτιστη μεταφορά στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Είναι πολύ σημαντικό όμως ε, να υπάρχει μια διατροπική προσέγγιση και μέσα σε αυτή να αναγνωριστεί πλήρως η συνεισφορά της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μια συστηματική ολοκλήρωση και ενσωμάτωση των στόχων του ΝΑΙΑΔΕΣ 2 είναι αναγκαία έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι πολιτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, για παράδειγμα, πιστεύω ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θα πρέπει να αναγνωρίσει την ανάγκη δημιουργίας κατευθυντηρίων γραμμών οι οποίες θα είναι αναγκαίες για τη δημιουργία οποιασδήποτε νέας βελτιωμένης προσέγγισης. Θα ήθελα να εστιάσω καταρχάς στην υποδομή που πιστεύω πως είναι το πιο σημαντικό συστατικό στοιχείο του προγράμματος ΝΑΙΑΔΕΣ. Στη Λευκή Βίβλιο Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί του στόχους για την πιο αηφόρο εσωτερική μεταφορά. Η εσωτερική λιμένες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο μιας βιώσιμης μεταφοράς, διατροπικής μεταφοράς, διότι χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να έχουμε αυτήν την ε, πολυτροπικότητα. Το σημαντικό ζήτημα λοιπόν είναι πώς η εσωτερική λιμένες και η εσωτερική ναυσιπλοεία θα ενσωματωθεί στους νέους αυτούς ε, διαδρόμους. Οι ναϊάδες φτάνουν μέχρι ένα σημείο και μετά υπάρχουν ασάφειες. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να κοιτάξετε λίγο περισσότερο τις ε, λεπτομέρειες του πώς θα ενσωματωθούν οι εσωτερικοί λιμένες στο πρόγραμμα Ναϊάδας. Η νέα πολιτική TNT αναφέρεται σε εννέα διαδρόμους, κεντρικούς διαδρόμους του δικτύου. Θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο εργασίας το οποίο θα συμπεριλαμβάνει ε, αυτούς τους διαδρόμους, και θα είναι βασισμένο στην ανάλυση των πληροφοριών που έχουμε από τα εθνικά σχέδια υποδομών, από τα σιδηροδρομικά δίκτυα και τις εμπορευματικές μεταφορές. Και εδώ υπάρχει η πρόκληση, διότι οι διάδρομοι έχουν μεν έτοιμα τα σχέδια για την εφαρμογή τους, ε, όμως τέτοια σχέδια εφαρμογής δεν υπάρχουν κατά ανάγκη και για τους εσωτερικούς λιμένες και δεν συμπεριλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια υποδομών. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό στις γνώσεις μας ε, όσον αφορά τους εσωτερικούς λιμένες και χρειάζεται περαιτέρω σχεδιασμός και βελτιωμένος σχεδιασμός έτσι ώστε να ενσωματωθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο εσωτερικοί λιμένες στα διατροπικά δίκτυα. Υπάρχει μεν κάποιος σκελετός, είναι όμως λιγότερο λεπτομερής από όσο θα θέλαμε. Χρειάζεται ε, λοιπόν πιο προσεκτική ανάλυση των εσωτερικών ελλημένων και του σχέδιου για τους ε, διαδρόμους έτσι ώστε να ενσωματωθούν στο δίκτυο αυτό οι εσωτερικοί λιμένες είναι πάρα πολύ σημαντικοί, όπως είπα, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορεί να υπάρχει νέα προσέγγιση στο, ε, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και δεν θα μπορεί να υπάρξει ε, διατροπικότητα. Έπειτα, θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, ενσωμάτωση των εσωτερικών λιμένων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όπως ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ανακοίνωση για τις ε, νεάδες και στο πακέτο για την κινητικότητα, οι ε, πιλωτές οδοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν εμπορεύματα και αγαθά και έχουν ε, τεράστιο δυναμικό. Η καλύτερη εξοποίησή του όμως θα γίνει με την καλύτερη ενσωμάτωση των εσωτερικών λιμένων στο δίκτυο. Και εδώ θα ήθελα να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενσκύψει στο ζήτημα αυτό και να φροντίσει να δημιουργηθούν βελτιωμένα σχέδια κινητικότητας για, την, για τις ε, μεταφορές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που συνδέεται περισσότερο με το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε, την οικονομική υποστήριξη για την ε, την ανακαίνιση των σκαφών και τον εξυγχρονισμό τους. Αυτό θα βοηθήσει τον ε, τομέα να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του και να την αυξήσει. Ε, θα ήθελα να σας πω τέλος ότι η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει το πρόγραμμα Ναϊάδες, όμως χρειάζεται προσοχή για να μην καταλήξει να γίνει μία τίγρη χωρίς δόντια, όπως λέμε και στη Γερμανία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την ανακοίνωση και πιστεύω πως ε, με βάση αυτή θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και ενδεχομένως να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρτζεκ έχει το λόγο, Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής του Δούναβη. Έχετε το λόγο. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of... Καλημέρα κυρίε και κύριοι, εκ μέρου τη Επιτροπή του Δούναβη καλωσορίζω όλους συμμετέχοντε στη σημερινή εκδήλωση. The is... Η Επιτροπή του Δούναβη είναι από τι πιο παλιέ διακυβερνητικέ οργανώσει στην Ευρώπη και ο Δούναβης είναι ο πιο διεθνή ε, ποταμό και συνέβαρε τα μάλα στην εξέλιξη των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων στην Ευρώπη. Η παρούσα επιτροπή είναι διεθνής διακυβερνητική ε, οργάνωση, οργανισμός, η σύμβαση για το καθεστώς της ναυσιπλοείας στο Δούναβι, στη, της διάσκεψης του Βελιγραδίου του 1948 δημιούργησε την Επιτροπή του Δούναβι. Η Επιτροπή έχει 11 κράτη-μέλη, 7 από αυτά είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε 9 χώρες παρατηρητές, 6 από αυτές είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα καθήκοντα της ε, Επιτροπής τη Σύμβαση, όπω αναφέρει στο άρθρο 8 τη Σύμβαση του Βελιγραδίου, όπω υποχρεωμένοι να καθορίσουμε τα διάφορα μέτρα για το Δούναβι προ όφελο ναυσιπλοεία. Χρειαζόμαστε επίση να έχουμε ένα ενοποιημένο σύστημα σημάτων και υπηρεσιών πλοήγηση και να έχουμε επίση κανόνε κοινού για την υποπτήρια των ποταμών. Χρειαζόμαστε επίση να παρέχουμε υδρομετεωρολογικέ υπηρεσίε, εναρμόνιση των κανόνων εσωτερική ναυσιπλοεία, να δίνουμε συμβουλέ και συστάσει, να δίνουμε στατιστικά στοιχεία στον αφορά την ναυσιπλοεία στο Δούναβι και να, κάνουμε, να εκδίδουμε δημοσιεύσει και τεχνικέ προδιαγραφέ. Αυτέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Ασχολούμαστε με αυτέ, ασχολούμαστε με τι υποδομέ και είμαστε έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δήλωση του Λουξεμβούργου όσον αφορά τις αποτελεσματικές υποδομές ε, των οδών ε, εσωτερικής αυσοπλοείας και τη συντήρηση του Δούναβη και των ε, διαφόρων παραποτάμων είναι κάτι που εγγράφει κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η δήλωση υπεγράφει από τις περισσότερους υπουργούς των χωρών που συμμετέχουν στην υπηρεσία και ανακρίθησαν και από την Σερβία και τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Σύμφωνα με τη δήλωση, η εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται πρέπει να ελέγχονται τακτικά και πρέπει να υπάρχει και ο μηχανισμός υποβολής εκθέσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη. Και θα υπάρχει και συντονισμός με την Επιτροπή του Δούναβη. Υπάρχουν επίγουσε ανάγκε στο Δούναβη, όπως προβλήματα που αφορούν την υλοποίηση των αρχών τη δήλωση και τη λύση προβλημάτων. Το TNT και το CF τα δύο αυτά προγράμματα θα συμβάλλουν τα μάλα στην ε, επίλυση των προβλημάτων. Βλέπετε στη διαφάνεια το σχέδιο δραστηριοτήτων για φέτος. Πρώτα απ' όλα έχουμε συνεδρίαση με τους γενικούς διευθύντες, ε, διευθυντές διαφόρων ε, εταιριών ναυσιπλοείας, μεταφορών. Ο τομέας θα μας δώσει πληροφορίες, πολύ σημαντικό για μας. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Move, και θα παίξουμε το ρόλο συντονιστή για την συντήρηση του Δούναβη ως διόδου μεταφοράς. Θέλουμε να έχουμε συμμαχία και συνεργασία με τις αγορές, με άλλες αγορές της περιοχής του Δούναβη, της ευρύτερης, της λεκάνης της περιοχής του Δούναβη και θέλουμε να συνεργόμαστε με το CSNR όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς. Έχουμε δύο νέα προγράμματα με το CSNR. Έχω, ετοιμάζουμε ένα γλωσσάρι για την εσωτερική ναυσιπλοεία και θα έχουμε κοινή ε, ορολογία που χρησιμοποιούμε τη εσωτερική ναυσιπλοεία και θέλουμε να οργανώσουμε και εργαστήριο, σεμινάριο για ε, την ε, ναυσιπλοεία αναψυχής. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να διοργανώσουμε συνεδρίαση που θα ακολουθήσει τη δήλωση του Λουξεμβούργου. Η συνάντηση να είναι υπουργικού επίπεδου. Έχει προγραμματιστεί να γίνει ε, αργότερα, τέλος Ιουνίου. Γιατί θέλουμε τη διοργάνωση συνεδριάσεως, διότι από το 2012, Ιούνιο 2012, δεν έγινε τίποτα όσον αφορά το Δούναβι και τις υποδομές του ή δεν έγιναν πολλά πράγματα τουλάχιστον. Θέλουμε να συμμετάσχουμε και στον ΑΙΑΔΕΣ 2 και στο ΣΕΣΤΕ. Όσον αφορά τον ΑΙΑΔΕΣ 2, η Επιτροπή του Δούναβι υποστηρίζει την αρχή της ποιότητας εσωτερικής αυσιπλοείας και το επίπεδο, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής ε, Υπήρου και υποστηρίζουμε την αρχή της πράσινης προσέγγισης και της καινοτομίας. Όσον αφορά το επταετές ε, πρόγραμμα, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τις τεχνικές απαιτήσει. Υποστηρίζουμε την ιδέα που έχει υποβληθεί για πανευρωπαϊκές προδιαγραφές υπό την προϋπόθεση ότι η άποψη όλων των κρατών μελών του Συμβουλίου του Δούναβη, της Επιτροπής του Δούναβη θα λαμβάνονται υπόψη. Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράσει υποστήριξη για την εσωτερική ναυσιπλοεία και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της οικονομικής κρίσης του τομέα και της ε, ε, πλοησιμότητας ε, των εσωτερικών αυτών οδών, πλωτών οδών. Υπάρχει κρίση στις περισσότερες χώρες, τις παραδουνάβιες. Τα τελευταία 20 χρόνια κατασκευάσαμε μόνο ένα φορτηγό πλοίο στο Δούναβι. Τα τελευταία 20 χρόνια κατασκευάστηκε μόνο ένα πλοίο. Όσον αφορά τις πληροφορίες που διαθέτουμε, δεν υπάρχει κάποια εταιρεία τα τελευταία χρόνια μεταφοράς, ε, ναυτιλιακή εταιρεία που να έχει κάνει ε, κέρδη τα τελευταία πέντε χρόνια. Να στείλω ένα μήνυμα τέλο προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή του Δούναβη θα υποστηρίξει μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση για την εσωτερική ναυσιπλοεία και κλείνω λέγοντα τα εξή. Res non verba. Θέλουμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι δεν μπορούμε, ο χρόνο δεν μα επιτρέπει να διαμαρτυρόμεθα. Πρέπει να δράσουμε, να εφαρμόσουμε υφιστάμενου μηχανισμού να λειτουργήσουν, όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμμετάσχουν στι συζητήσει και να βρούμε νέες κατευθύνσεις για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Αυτά και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πετάρ, επόμενος. ETF. Ο Γενικός Γραμματέας του Nautilus International ε, εκπροσωπεί τη Διεθνή Οργάνωση των Εργαζομένων στον τομέα. gelegenheid biedt om het thema van vandaag, towards an optimal integration. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε ως εκπρόσωπο των συνδικάτων για αυτό το θέμα, την οργάνωση δηλαδή των εσωτερικών πλωτών οδών ε, και των ΑΙΑΔΕΣ 2, ώστε να σας δώσω την γνώμη των συνδικάτων. Τι σχέση έχουν τα συνδικάτα, θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, ε, εφόσον εμείς περιοριζόμαστε στη κοινωνικά θέματα και στη εξασφάλιση των θέσεων απασχόλησης. Όμως αυτό δεν αληθεύει ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Ε, Ευρωπαϊκό Συνδικάτο, ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και ότι μπορεί να υπάρξουν καταχρήσεις έναντι των εργαζομένων. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα η συνέπεια των μεγαλύτερων πιέσεων διαρκώς και θα πρέπει να δείχνει κανείς πολύ καλή θέληση. Ποιοι είναι τώρα οι εξωτερικοί παράγοντες. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα ε, ε, από το λιμάνι του Ρότερνταμ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των μεγάλων προγραμμάτων υποδομών, για παράδειγμα για το δεύτερο τέρμιναλ του Ρότερνταμ, όλες οι αρχές, ε, οι λιμενικές, αλλά και οι φορείς δεν έλαβαν υπόψη τις συνέπειες ε, ε, της της παρουσίας, της, της οργάνωσης μάλλον της επιμελητίας στην ξηρά. δεν έλαβαν υπόψη τη γνώμη δηλαδή των ε, συνδικάτων ε, στην ε, οργάνωση επιξήρας. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα λήφθη όμως υπόψη η γνώμη των εφοπλιστών. Θα πρέπει να βλέπουμε την, το εύρος των του βυθίσματος, ε, τις ε, λεκάνες ε, στάθμευσης των σκαφών και ούτω καθεξής. Επίσης υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την, τον ελιμενισμό των πλοίων. Δηλαδή έγινε περισσότερη μελέτη στη θάλασσα παρά στην ξηρά. Οι εφοπλιστές δεν ενδιαφέρονται για τη σωστή διαχείριση στη ξηρά. Ε, έχουν ε, ποσοστά ε, που ελέγχονται από τους ίδιους, γύρω στο 30% και από τη στιγμή που τα κοντέινερ βγαίνουν στη ξηρά και μπαίνουν πάνω στις παλέτες, τέρμα τα έξοδα για τους εφοπλιστές. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει. Μετά είναι ο διανομέας που έχει, φέρει την ευθύνη. Είναι οι μεταφορικές εταιρείες που ασχολούνται με τη μεταφορά όλων αυτών των εμπορευματοκιβωτίων. Μόνο λοιπόν η θαλάσσια μεταφορά ε, που φέρει έσοδα στα λιμάνια και η εσωτερική πλοήγηση, ναυσιπλοεία θεωρείται επιπλέον κόστος και πόρος Ποιες είναι λοιπόν οι συνέπειες όσον αφορά την εσωτερική ναυσιπλοεία στο θέση της εσωτερήκευσης των δραστηριοτήτων, το Ρότερνταμ δυστυχώς επέλεξε την αποκέντρωση των σταθμών, των τέρμιναλ. Αντί να υπάρχει ένα σημείο ε, φόρτωσης-εκφόρτωσης, υπάρχουν 7 ή 8. Και αυτό ισχύει και για τα εμπορεύματα στο Terminal 1, στο Terminal 2. Αυτό επιφέρει καθυστερήσεις, αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό φαινόμενο. Μετά από την αποκέντρωση, οι ιδιοκτήτες, οι πλειοκτήτες, δεν ασχολούνται πλέον με την εκφόρτωση των εμπορευμάτων. Ένα σύντομο παράδειγμα. Ένα εμπαρομετοκιβώτιο ξεφορτώνεται στην ξηρά και μετά πρέπει να μετακινηθεί από το ένα τέρμιναλ στο άλλο. Από κάποιον φορέα εσωτερικής ναυσιπλοείας. Όπως το ECT. Αυτό βεβαίως οδηγεί σε καθυστερήσεις και αυξάνεται ο χρόνος παραμονής των ε, κοντέινερ στο λιμάνι και δημιουργείται συμφόρηση, αλλά και αύξηση του κόστους και για τους φορείς της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Οπότε η τοπική και η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν ώστε να αποφευχθεί ο κορεσμός, η συμφόρηση αλλά και για να ε, βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της εσωτερικής ταυσιπλοείας η οποία έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτής της υποτιθέμενης βελτιστοποίησης και Βεβαίως ε, πρόκειται για αύξηση του κόστους των μεταφορών που με τη σειρά του μεταφράζεται σε αύξηση του γενικού κόστους ε, με ό,τι αυτό επιφέρει, ε, συνεπάγεται. Εμεί θα θέλαμε να υπάρχει ένας οικονομικός μηχανισμός ώστε να αποφεύγεται το κοινωνικό dumping όσον αφορά τους εργαζόμενους διότι υπάρχει διαρκώ περισσότερη πίεση για την μείωση του κόστου ε, στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Αν οι πλειοκτήτε και οι λιμενικέ αρχέ δεν έχουν κανένα οικονομικό πλονέκτημα από την οργάνωση τη εσωτερική ναυσιπλοεία και εξακολουθούν να τη θεωρούν ω απλώ ένα επιπλέον κόστο, δεν θα μπορέσει να υπάρξει μια βέλτιστη ολοκλήρωση τη εσωτερική ναυσιπλοεία στο πλαίσιο μια ε, ε, ολοκληρωμένη αλυσίδα επιμελητία και υποδομών. Εμεί γνωρίζουμε γνωρίζουμε πώς το πρέπει να λύσει αυτά τα προβλήματα. Για παράδειγμα υπάρχει το πρόγραμμα Logic, το σχέδιο Logic. Ωστόσο, ακόμα διερωτώμαθα αν θα καταστεί δυνατή η ε, ε, ολοκλήρωση. Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν λαμβάνεται δε υπόψη καθόλου. Εμείς τα συνδικάτα ζητάμε την εκπόνηση ε, υποδομών, προγραμμάτων υποδομών, όπως αυτό το Logic, ε, που θα λαμβάνει υπόψη το παράγοντα του ανθρωπίνου δυναμικού. δυναμικού με συγχωρείτε. Και θα θέλαμε να δούμε αν υπάρχει κάποια δυνατότητα βοήθειας για αυτά από την ευρωπαϊκή πλευρά. Τελειώσαμε το πρώτο πάνελ. Κυρία Μάστινερ και ο κύριος Βαντάλεν από τα μέλη θα να πάρουν το λόγο. Άλλος της. Ε, ξεκινάμε από σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν περίμενα να μιλήσω πρώτη. Έχω ορισμένε ερωτήσει για όλου του ομιλητέ. Καταρχά, να σα ευχαριστήσω όλου ε, που ήρθατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσε οι εισηγήσει σα. Καταρχά, ε, κυρία Τεσλέπερ, είπατε πολύ καλά λόγια για το ΤΕΝΤΕ και συμφωνώ μαζί σα. Είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν και τα δύο προγράμματα. Και όντω οι εσωτερικέ πλωτέ οδοί παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μας αναφέρατε τα σημαντικά λοιπόν σημεία. Τώρα κύριε Στάκα, ε, μου άρεσε πάρα πολύ η εισήγησή σα. Μου άρεσε πάρα πολύ το επιχείρημά σα ότι είναι πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο των ε, διατροπικών μεταφορών οι εσωτερικέ πλωτέ οδοί και πραγματικά είναι, ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον. το πόσο σημαντικέ είναι αυτέ με τα παραδείγματα που μα δώσατε για το Τούσπρο και και το Ρήνο. Μία ερώτηση στο Κοινοβούλιο είχαμε μία ακρόαση για το λιώσιμο των επαγετώνων και την άνοδο της στάθμης των εσωτερικών πλωτών οδών. Θα ήθελα ε, να σας ερωτήσω αν έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό και ποια θα ήταν η αντίδρασή σας σε μια τέτοια περίπτωση. Τώρα, κυρία Όμπστ, είπατε ότι θα επιθυμούσατε να συνδέονται καλύτερα οι εσωτερικοί λιμένες με τα ε, αστικά κέντρα και έτσι ώστε να βελτιωθεί η κινητικότητα. Μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν ήδη υποδομές και ότι μπορούν αυτές να βελτιωθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, ε, κύριε Μάργιτς αναφέρεται πως ε, υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί μία ενιαία ορολογία στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Ε, και θα ήθελα να πω ότι καταρχάς συμφωνώ μαζί σας, αλλά ποια γλώσσα θα επιλέξουμε για την ε, ορολογία αυτή, διότι θα επικρατήσουν τα αγγλικά, γιατί όχι και μια άλλη γλώσσα. Τώρα, ε, αναφέρθηκε και επίσης ε, αναφερθήκατε επίσης για την ε, ελκυστικότητα του επαγγέλματος, για το πώς θα κάνουμε ε, το επάγγελμα της αστυνομικής ναυσιπλοείας σε πιο ελκυστικό και ίσως και όχι μόνο για τους άντρες. Ίσως εσείς θα μπορούσατε να μας αναφέρατε ορισμένες προτάσεις σας γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε κύριος Βαντάλεν. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ε, σημερινή ακρόαση. Ακούσαμε τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις οποίες θα τις συζητήσουμε. Οι εσωτερικές πλωτές ε, οδοί όμως είναι πολλά περισσότερα από δύο απλές προτάσεις. Και αυτό φαίνεται βλέποντας και την νομοθεσία. Είναι προφανές ότι χρειάζεται να συζητήσουμε περισσότερο το ζήτημα των εσωτερικών πλωτών οδών, διότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και άμεσα συνδεδεμένο με την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Στάκερ και τον κύριο Μάρτσιτς. Όσον αφορά τις ε, υποδομές, η κυρία Μάισνερ αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα επίσης. Ακούτε υπέροχες ιστορίες που λέγονται για τις υποδομές και πόσο σημαντικές είναι. Αλλά πολλές φορές έχουμε συμφορήσεις. Εμπλοκή της κυκλοφορίας στην ε, Ευρώπη. Συζητήσατε με τη νέα κυβέρνηση Μέρκελ για να θέσετε αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν διάφοροι τομείς που θα πρέπει να εξεταστούν, Ούτως ώστε να συντηρείται σωστό επίπεδο η στάθμη των υδάτων. Για να έχουμε το σωστό επίπεδο ε, για πάνω από 300 μέρες το χρόνο. Δεν θέλουμε να φύγει η κυρία Μέρκελ χωρίς να γίνει τίποτα. Θα πρέπει ε, στις δεξαμενές να φροντίζουμε να υπάρχουν αρκετά αποθέματα για να συμπληρώνουμε. Όταν κατεβαίνει η στάθμη, συμπληρώνουμε τη στάθμη του νερού. Για να υπάρχει δυνατότητα ναυσιπλοείας. Κάτι άλλο. Δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά το θέμα αυτό. Για τους διαδρόμους κάναμε, για τους διαδρόμους μεταφορών κάναμε κάποια πράγματα. Θα ήθελα περισσότερα να γίνουν όμως όσον αφορά το συντονισμό των δυνάμεων. Όλοι να ξέρουν τι πρέπει να γίνει. Ε, νομίζω ότι είναι μετριοπαθής η προσέγγιση σας. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες πρωτοβουλίες. Να συζητήσουμε, θα μπορούμε να συζητάμε θεωρητικά για τις υποδομές ε, ε, ε, για για πάντα. Αν δεν κάνουμε κάτι όμως θα μείνει έτσι η κατάσταση. Λοιπόν, αναφερθήκατε στην καινοτομία, ότι είναι αναγκαία καινοτομία. Αναφέρθηκε από κάποιον συνάδελφο. Ναι, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αλλά είναι ένας αόριστος στόχος, ανοιχτός στόχος. Όλοι θα συμφωνήσουν. Αλλά όχι όλες οι καινοτόμες ιδέες είναι χρήσιμες. και τα καινοτόμα άτομα είναι σημαντικό να συνεργαστούν. Αλλά ε, η συνεργασία μεταξύ πλειοκτητών και αυτοκινητοβιομηχανίας, η συνεργασία με τους σιδηροδρόμους, μια σύμπραξη. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει καινοτομία. Έχουμε μεγάλο κατακαιρματισμό. Μπορείτε να δεχτείτε αυτού του τύπου την καινοτομία όσον αφορά τη συνεργασία των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και των διαφόρων φορέων ε, θέλατε να προωθήσετε ε, τα διάφορα είδη μεταφορών. Τι κάνει ο τομέας. Μιλάμε για υποστήριξη, μιλάμε για χρήματα γενικά. Ο τομέας ο ίδιος αυτός τι κάνει. Τι κάνει για να εξασφαλίσει ότι ε, οι διάφοροι τρόποι μεταφορών ε, δίνουν θέμενη αξία και να το εκτιμούν οι διάφοροι αυτό. Επόμενος. Κύριος Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονε για τη σημερινή ακρόαση. Είναι πραγματικά απόλυτα αναγκαίο όταν αναφερόμαστε στην ε, ενίσχυση Τη εσωτερική ε, ναυσιπλοεία ε, στην Ευρώπη, τη ναυσιπλοεία, να ε, δούμε ιδιαίτερα το θέμα των εσωτερικών λιμένων, διότι ο τομέας αυτός έχει το χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα, καταναλώνει την λιγότερη ενέργεια. Όμως, Υπάρχει μεγάλος δισταγμός, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την εσωτερική ναυσιπλοεία, λόγω του περιβάλλοντος. Αναφέρεται πολύ συχνά η περιβαλλοντική καταστροφή, η άνοδος της ε, στάθμης, των ποταμών, ε, του, Έλβα, του Ρήνου. Και πραγματικά υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει πρόβλημα, για παράδειγμα, στο... Ε, συμφόρηση στη σύνδεση Ρήνου και Δούναβη. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και ιδιαίτερα μεταξύ Ρήνου και Δούναβη δεν υπάρχει κάποια ε, λύση προς το παρόν. Το πρόγραμμα Ναϊάδες είναι ένα γενικότερο πρόγραμμα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά επιμέρους ε, λιμάνια, δικτύωση, αλλά πρέπει πιστεύω να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι υλοποιήσιμο και θα έχει αποτελέσματα, να μην κατακαιρματιζόμαστε παντού. Υπάρχουν κάποια σχέδια στη Γερμανία για τη σύνδεση του καναλιού Ερίνου και Δούναβη. Φυσικά υπάρχουν και εσωτερικές αντιθέσεις ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατήδια. Αυτό όμως δείχνει πόσο αναγκαίο είναι οι εσωτερικοί λιμένες να πιστοποιηθούν και να γίνουν και να αναγνωριστεί η αξία τους ως κομβικά σημεία, ως κομβικοί λιμένες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υποδομή της Ευρώπης αυτό. χρειάζεται σχεδιασμός, σωστός σχεδιασμός για την διεύρυνση της χωρητικότητας και αυτό χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό όχι μόνο λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση αλλά και την υποδομή και το μέλλον της, των μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες και όσους διοργάνωσαν την ακρόαση. Είναι ένα θέμα ενδιαφέρον που μένει στο περιθώριο. Έχω δύο εκπλήξεις όμως να εκφράσω. Εκφράστηκε, αναφέρθηκε μια ε, έρημνα για να γίνει η αναβάθμιση των σκαφών όσον αφορά το θόρυβο των κινητήρων και γενικά των σκαφών. Άκουσα αυτό το retrofitting. Δράτω με τη ευκαιρία να πω ότι απ' την άλλη υπάρχει κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό και δεν εκφράστηκε ξεκάθαρα από τους συμμετέχοντες. Η τυποποίηση είναι αυτό το θέμα και των σκαφών ανάλογα με το μέγεθος και του υλικού που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων, φορτοεκφόρτωση κλπ. Έχουμε εμπορευματοκιβώτια που πάνε στα πλοία. Μιλάμε για εσωτερική ναυσιπλοεία και δεν αναφέρονται αυτά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται. Ε, ποια είναι τα, τα στα πλοία, τύπος εμπορευματοκιβωτίων, γερανογέφυρες κλπ. Αυτά δεν αναφέρθηκαν λεπτομέρως. Με έκπληξη άκουσα όσον αφορά το λιμάνι του Ρότερνταμ κάτι. Είναι το πρώτο στην Ευρώπη και ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα θέσεων. Κυρίως όσον αφορά τα φορτία πάνε στην οδοχώρα. Ε, υπάρχει έλλειψη διασύνδεσης για να υπάρχει σωστή διασύνδεση ε, μεταξύ των εμπορευμάτων που φτιάχνουν από τη θάλασσα και πώς μεταφέρονται μετά στους άλλους τρόπους μεταφοράς από τη ξηρά. Είναι σημαντικό το το λιμάνι και όχι μόνο για τη Βόρεια Θάλασσα. Υπάρχουν προτάσεις όσον αφορά τη λειτουργία του λιμανιού να βελτιωθεί. Ε, ρωτάω την, Ευρω... την Επιτροπή. Μπορούμε να δράσουμε, να κάνουμε κάτι Και κάτι άλλο που θέλω την άποψη των μελών του πάνελ. Στο Κοινοβούλιο υποστηρίξαμε την προσέγγιση για την ο, το να ενταχθούν στους διάφορους διαδρόμους ε, τα διάφορα ποτάμια και παραπόταμοι, οι δύο διεσωτερικής ναυσιπλοείας. Το ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το στήριξε το Συμβούλιο, καταφέραμε το εισαγωγικών να βάλουμε έξι ε, ποταμούς σε αυτούς τους διαδρόμους μεταφορών. Κάτι που δεν αναφέρεται όμως είναι το σύνολο των... Να, είναι, υπάρχει, να θεωρείται ευρωπαϊκό σύνολο, ενιαίο το σύστημα των ε, ευρωπαϊκών ε, ποταμών. Άκουσα να αναφέρεται ο Δούναβης, η διασύνδεση μεταξύ Ρήνου και Δούναβη. Δεν μιλήσατε όμως, ή δεν άκουσα εδώ, να μιλήσετε για άλλες διασυνδέσεις τι γίνεται, πώς συνδέονται οι διάφορα ποτάμια με το Ρήνο και το Δούναβι. Δηλαδή όλο το σύστημα, το ποτάμιο, ε, το, να διασυνδέεται στην Ευρώπη. Να δημιουργεί ένα νέο σύνολο. Δηλαδή είναι σαν να εξετάζουμε διάφορα κομματάκια, ε, ε ανάντι και κατάντι του Δούναβη κλπ, ε, κομμάτια του Ρήνου, καθένας ασχολείται με το μικρό του κομμάτι και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη γενική σφαιρική προσέγγιση. Δεν άκουσα εκείνοι που ασχολούνται με το Δούναβι μαζί με, την, ε, με τον Φορέκ Μετάδευσης του Ρήνου να μιλήσουν για διασυνδέσεις, κοινά προγράμματα κλπ. Εδώ δεν άκουσα. Μπορεί να υπάρχουν τέτοια προγράμματα, εδώ δεν άκουσα να αναφέρεται κάτι τέτοιο. Τέλος, σε ποια δεδομένη στιγμή θα υπάρχει αρχή που θα ασχοληθεί με όλο το σύστημα. ένας φορέας που θα ασχοληθεί με όλο το ποτάμιο σύστημα. Αυτό καθ' αυτό, σαν ένα σύνολο συνεκτικό. Και πότε θα σταματήσουμε να κατακαιρματίζουμε το ποτάμιο σύστημα. Το σύνολο των υποδομών, σαν, μια λεκάνη ε, ε, με την, και να ασχολούμαστε με την διοργάνωση όλη αυτής της κοινή ε, λεκάνης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που διοργάνωσαν αυτή την ακρόαση, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα πρόταση που μας υπευλήθη. Το ΝΑΙΑΔΕΣ 2 είναι σημαντικότατο πρόγραμμα για τις ευρωπαϊκές μεταφορές και γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω τη σύμφωνη γνώμη μου όσον αφορά αυτά που είπε τώρα ο Ντομινίκ. Δηλαδή, Κρίμα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε μια κοινή στρατηγική, ενιαία στρατηγική για τα εσωτερικά ποτάμια. Μια συνεκτική στρατηγική που να μπορεί να μην εξετάζει μόνο τις μεταφορές μέσω ποταμών, την ανάπτυξη των στόλων και των εσωτερικών ε, λιμένων, αλλά και τις πτυχές που αφορούν το περιβάλλον, την περιφερειακή ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη. Όσον αφορά το Δούναβι, εγώ γεννήθηκα σε μια πόλη που βρίσκεται ε, στις όχθες του Δούναβι. Και βέβαια ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο ε, αναπτύσσεται και θα αναπτυχθεί ο Δούναβης και μεταφορέ το στο Δούναβη στο μέλλον. Μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη, η σύνδεση του Δούναβι με τους άλλους ποταμούς. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να αμελείται. Υπάρχουν κάποιοι που είναι κατά αυτής της διασύνδεσης. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι οι πλειοκτήτες θα μπορούσαν να μειώσουν τις τιμές, να μειωθεί το κόστος, θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε ένα τμήμα της αγοράς. Ε, δεν συμφωνώ με αυτό. Πρέπει να έχουμε μια αγορά εσωτερική και είναι σημαντικό για την Ευρώπη να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ ε, Ρήνου, Δούναβη, ε, Ευξήνου Πόντου κλπ. Όσον αφορά την ανάπτυξη των οδών αυτών, των διαδρόμων, πρέπει να βελτιώσουμε τα λιμάνια. Στη Ρουμανία δυστυχώς τα τελευταία 20 χρόνια οι επενδύσεις ήταν ελάχιστες όσον αφορά την ανάπτυξη των λιμένων και των διαφόρων ε, ποταμίων διαδρόμων. Και γι' αυτό ο μηχανισμός αυτός που αφορά τη διασύνδεση, τη σύνδεση των διαφόρων σημείων της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικός. Ποιε είναι οι συνθήκες όμως για τη χρηματοδότηση, για πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αναφέρθηκα στον εξυγχρονισμό των ε, στόλων. Διαμαρτύρονται οι πλειοκτήτες διότι λένε ότι οι συνθήκες για την πρόσβαση στους πόρους είναι ε, πάρα πολύ δύσκολες, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και εξαιτία αυτού υπάρχουν πολλοί πλειοκτήτες που δεν θέλουν καν να ζητήσουν ε, να αποκτήσουν αυτούς τους πόρους. Και γι' αυτό πιστεύω ότι εμείς που ασχολούμαστε με την νομοθεσία, που είμαστε υπεύθυνοι για τέσπιση νομοθεσίας, πρέπει να φροντίσουμε ότι ώστε οι συνθήκες για την χρηματοδότηση στα πλαίσια του ΝΑΙΑΔΕΣ 2 να είναι η απλούστερη δυνατή. Ε, χρειαζόμαστε συνεχή διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εμπλεκομένων φορέων, εκείνων που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα ΝΑΕΑΔΕΣ 2. Ούτως ώστε αυτές οι συνθήκες για τη χρηματοδότηση να προσαρμοστούν σωστά, να είναι απλοί οι κανόνες. Δεν θέλουμε κατάσταση παρόμοια με την κατάσταση που επικρατεί στο πρόγραμμα Μάρκο Πόλο. Υπήρχε ένα προπολογισμό, αλλά δυστυχώ τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε ο προπολογισμό. Γιατί? Διότι οι συνθήκε για την πρόσφαση του προπολογισμό ήταν πάρα πολύ ε, αυστηρέ. Και τέλο, η... Ε, αυτά ήθελα να πω. Και τελικά ότι δεν συμμετείχαν πολύ στο πρόγραμμα Μάρκο Πόλο για αυτό το λόγο. Ευχαριστώ από την πλευρά μου. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν είδατε τα Χριστούγεννα στο Ηνωμένο Βασίλειο το Discovery είχε ένα πρόγραμμα υπέροχο και ήταν ε, με τίτλο «Ο Δούναβης, ο Άγριος Δούναβης», «Wild Danube». Υπέροχο πρόγραμμα στο Discovery έδειχνε όλο το Δούναβη από Γερμανία μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, τον έξινο πόντο και έβλεπε το Δούναβη σαν ποτάμι. Υπέροχο πρόγραμμα ήταν. Τέλος πάντων, για να το ξέρετε σας το λέω. Γιατί είδα το πρόγραμμα. Διότι όλοι ερωτευτήκαμε το Δούναβι σε αυτή την επιτροπή. Σχετίστε με τη Σίλβια. Βέβαια είναι σαν υιοθετημένος μας ποταμός ο Δούναβης. Με κάθε σεβασμό προς το Ρήνο. Αλλά ο Δούναβης είναι το αγαπημένο μας ποτάμι. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι ερχόμαστε σε αυτό που ο Πίτερ Βαντάλεν είπε. Ο Ντόμινικ Ρίκε και όλοι έφυξαν και η Σίλβια κλπ υπάρχει έλλειψη κοινή προσέγγισης όσον αφορά τις εσωτερικές οδούς ε, ναυσιπλοείας. Η κοινότητα αυτή του τομέα δεν είναι ενοποιημένη. Όχι μόνο για να συνδεθούν μεταξύ τους, αλλά να συνδεθούν και με άλλους τρόπους μεταφορών. Να, εξεταστεί, να εξεταστούν υποδομές στο σύνολό τους. Η εσωτερική ναυσιπλοεία, οι εσωτερικέ οδοί είναι απόσπαστο τμήμα του αλυσίδα τη επιμελητία. Σωστά το βλέπουμε έτσι. Και σωστά δίνουμε προτεραιότητα στι εσωτερικέ οδού ναυσιπλοεία από αυτή την πλευρά. Αλλά είναι ευρύτερο το θέμα. Αφορά και άλλε υποδομέ. Δηλαδή, κατά πόσο οι δεξαμενέ χρησιμοποιούνται σωστά για να βελτιώνουν τη στάθμη των ποταμών κλπ. Έχω παράδειγμα από τη χώρα μου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ξέρετε ότι δεν έχουμε υπέροχε εσωτερικέ οδού ναυσιπλοεία. Έχουμε κάποια κανάλια πολύ στενά για τους τουρίστε. Υπάρχει μια εσωτερική οδό που χρησιμοποιείται εμπορικά. Το κανάλι του Μάντσεστερ και περνάει την περιοχή μου. Και θέλουμε να το αναπτύξουμε αυτό για να περνάει περισσότερη κυκλοφορία από τη θάλασσα της Ιρλανδίας και να φτάνει στο Μάντσεστερ. Υπέροχα. Ο ανοιχτός στόχος που ανέφερε ο Πίτερ αλλά ε, και τελικά είναι ελεύθερο χωρίς τερματοφύλακα το τέρμα και πρέπει να σας πω ότι ασχολούμαι με τα θετικά και πολύ συχνά πάνω σουτάρουν σε άδειο τέρμα και χάνουν και εδώ έχουμε ένα στόχο και το χάνουμε. Καλή ιδέα αυτή για να ανοίξει το κανάλι του Manchester αλλά κανείς δεν είδε ότι σε αυτό το κανάλι υπάρχουν δύο γέφυρες που ανοίγουν στο Warrington. Και αυτές οι δύο γέφυρες που ανοίγουν στο Warrington φέρνουν τις δύο αρτηρίες στο Warrington. Όταν έρχεται λοιπόν στο κανάλι του Manchester για να πάει στο Manchester ή να πάει από την άλλη πλευρά να πάει στο Liverpool ανοίγουν αυτές τις γέφυρες, τις πόρτες, αποτέλεσμα είναι κυκλοφοριακό house στο Warrington. Διότι κανείς δεν σκέφτηκε ότι αν βάλουμε περισσότερη κυκλοφορία στο κανάλι του Manchester πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης. Να είναι ένα πρακτικό παράδειγμα για την έλλειψη κοινή προσέγγισης αντιμετώπισης, κοινού προβληματισμού όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω. Πέτερ. Είναι αγαπημένο μας ποτάμι, όπως είπαμε, Πέτερο, Πέτερο Δούναβης. Και είπατε, η προησιμότητα του Δούναβη είναι ένα ζήτημα. Και συναφή ζητήματα που περνάει το ποτάμι από τη Σερβία και είπες ότι συμφωνείς με τις Ναϊάδες και είπες μια φρασούλα που νομίζα ότι μου θύμισε το πακέτο σιδηροδρόμων και είπες από τη στιγμή που όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν με αυτό είπες και αμέσως μπαμ τριν, χτύπησε ο συναγερμός τριν, τριν, τριν διότι να καταφέρεις να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη, ε, να συμφωνήσουμε σε κάτι δεν είναι κάτι εύκολο, το ξέρεις αυτό. Κυρίως όταν έχεις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί εντάσσεται ο Δούναβης. Τι γίνεται λοιπόν με την πλησιμότητα του Δούναβη. Διότι ε, πάει οπλοπλοίσιμο, εκεί από εδώ περνάει πλοίο, από εκεί δεν περνάει, αλλάζει ο Δούναβης. Ίσως να περνάει πλοίο από εκεί. Και δεν, γίνεται αυτό. Πώς να έχουμε έτσι ολοκληρωμένη εσωτερική ναυσιπλοεία, ένα σύστημα που θέλουμε. Καταλαβαίνω, όλα για χρήμα είναι, περί χρήματος πρόκειται, ποτέ δεν αρκούν τα χρήματα. Υπάρχουν αρκετά χρήματα για να πούμε την αλήθεια, αλλά πάντα σε λάθος χέρια. Αλλά ποτέ δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για να γίνουν αυτά. Και εδώ γίνεται μια προσπάθεια να ξεκινήσουμε τουλάχιστον να διοχετεύουμε, συγγνώμη για το αστιακή, διοχετεύουμε στο κανάλι, να ρίξουμε στο κανάλι χρήματα για να γίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα η ιστορική ναυσιπλοεία. Και συμφωνούμε όλοι με αυτό, κανείς εδώ δεν διαφωνεί. Δηλαδή αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να θέσουμε προτεραιότητες και να πάρουν μεγαλύτερη προτεραιότητα οι εσωτερικέ ε, οδοί ναυσιπλοεία, αλλά να συνδεθούν και με τα υπόλοιπα, του άλλου τρόπου μεταφορά. Καλά το είπε ο Ντομινίκ, να γίνει η διασύνδεση με τα άλλα ποτάμια, με το Ρήνο, ε, με όλα τα ποτάμια, το Λίγυρα κλπ. Μόνο το δίκτυο. Αυτά από πλευράς Προέδρου. Τρία λεπτά ο καθένας ένας ένας θα μιλήσετε, τα μέλη του πάνελ, αν μπορούσατε να περιοριστεί το καθένα σε τρία λεπτά. Κάρεν, Έρικ, Κάθλιν, Πέταρ, αυτή τη σειρά. Η Κάρεν ξεκινά πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα για το συνεκτικό αυτό σύστημα. Έχουμε μάλιστα και ένα χρονοδιάγραμμα πολύ συγκεκριμένο σχετικά με αυτό. Τώρα, για τα αγαπημένα project δεν μπορώ να πω ότι ισχύει κάτι τέτοιο λόγω αυτή τη συνεκτική άποψη. Τώρα, αν κοιτάξουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, θα δούμε ότι υπάρχουν ορισμένα προγράμματα τα οποία έχουν οριμάσει χρονικά και συνδέονται με αυτήν την συνεκτική προσέγγιση. Είναι έργα που είναι ήδη ενταγμένα, είναι όριμα. Αυτά λοιπόν ταιριάζουν με το πρόγραμμα αυτό και σίγουρα Εκεί δεν χρειαζόμαστε βοήθεια, τη δική σας βοήθεια. Έχουν ήδη υποβληθεί προτάσεις, ήδη δρομολογούνται τα έργα. Από την άλλη, υπάρχουν κάποια έργα τα οποία είναι υψηλή προτεραιότητα και δεν θα σα ε, ενοχλήσω πάλι να σα πω για το Straubing Hirschhofen, για το πρόγραμμα αυτό, αλλά τα προγράμματα αυτά είναι πολιτικά ευαίσθητα, υπάρχουν διαφωνίες ε, μεταξύ περιβάλλοντος και πλειοκτητών. Αυτό όμως στην ουσία δεν ισχύει. Και όταν οι δικοί προστρέχουν στις ε, κυβερνήσεις τους, ε, κοιτούς, κοιτούν αυτές τις τροπικότητες. Από τη μία έχουμε την εσωτερική ναυσιπλοή, από την άλλη το δικό δίκτυο, τους σιδηροδρόμους, τα οποία αυτά δίκτυα δεν μπορούν να ενωθούν και υπάρχουν διαφωνίες. Όμως εσείς ως ευρωβουλευτές έχετε και την ευρωπαϊκή διάσταση, άποψη και την τοπική της εκλογικής σας περιφέρειας. Ε, εσείς λοιπόν μπορείτε να βοηθήσετε έτσι ώστε να ξεπεραστούν αυτές οι διαφωνίες, αυτά τα εμπόδια. Και ο Έριχ το ανέφερε. Έχουμε αυτές τις ε, διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές τροπικότητες. Υπάρχουν οι εθνικές κυβερνήσεις, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτές οι διαφωνίες δημιουργούν το μεγάλο εμπόδιο. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαφορετικές απόψεις οι οποίες δυσχεραίνουν την ε, συνεκτική αυτή προσέγγιση, διότι μιλούμε αυτή τη στιγμή για μια αλυσίδα διακίνησης και μεταφοράς που πρέπει να ολοκληρωθεί. Το χρονοδιάγραμμά μας υλοποιείται μόνο μέσω ενός συνεκτικού και ποιοτικού συστήματος και πρέπει να φροντίσουμε ώστε να είναι υλοποιήσιμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στο στάδιο του σχεδιασμού να ληφθούν υπόψη και τα ε, τοπικά συμφέροντα και οι ιδιαιτερότητες, διότι εδώ υπάρχει η δυνατότητα για παράδειγμα της επέκτασης ενός λιμένα και να βγάλεις τα φορτηγά τα οποία διέρχονται από τις πόλεις. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων, για παράδειγμα, με την, ε, με την ε, ανάπτυξη, με τον χωροταξικό σχεδιασμό. για παράδειγμα, η περίπτωση του Σικουάνα. Ε, ο Σικουάνας ε, και οι γύρω περιοχές ε, είναι μνημείο πολιτισμικής εκκληρονομιά. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα και σπαταλάται πάρα πολύ χρόνο στον χωροταξικό σχεδιασμό έτσι, να μπορέσουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη όλες οι διαφορετικές συνιστώσεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν μέσω μια συνεκτική προσέγγιση και εσεί μπορείτε να παίξετε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και στην εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματο. Σα ευχαριστώ πολύ, Έρικ. Πιστεύω πω ε, πράγματι η παρατηρήσεις ήταν πολύ εύστοχες και όντως πιστεύω ότι η σύνδεση είναι η λέξη κλειδί. Δεν πρέπει να συνδεθούν μόνο οι εσωτερικές απλωτές οδοί μεταξύ του, αλλά και με τα οδικά δίκτυα και κυρίως με τους ε, με τους ε, παράγοντες, με τους ε, φορείς οι οποίοι χρησιμοποιούν τις οδούς αυτές και πρέπει να δούμε πραγματικά πώς θα υλοποιηθούν τα προγράμματα αυτά, με ποιο τρόπο. Και εδώ πέρα δεν αρκεί μόνο η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρειάζεται να συμπεριληφθούν όλες οι ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα, οι μεταφορικές και να δουν πραγματικά ότι είναι προς το συμφέρον τους η δημιουργία μιας ε, Βιώσιμε λύσει, διότι πραγματικά είναι και οικονομικά πιο βιώσιμη, όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να ε, χρειαστεί να δημιουργήσουμε προτεραιότητες, εκεί πρέπει να δούμε πραγματικά πώς έχουν τα πράγματα. Αναφερθήκατε και στον Μοζέλα. Ο Μοζέλα είναι ένας ποταμό με εκατομμύρια σε επενδύσεις. και σε επενδύσεις ακινήτων και αυτό έχει οδηγήσει σε διαφωνίες ως προς την χρήση του ως εσωτερική πλωτή οδό. Επίσης, αυτές οι προτάσεις και τα έργα που θα γίνουν θα πρέπει να γίνουν φυσικά με απόλυτη διαφάνεια. Τώρα, ρωτήσατε τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Πολλά κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Πριν από 15 χρόνια ήμουν ε, στην ομάδα που δημιούργησε έναν ε, τοπικό, ένα τοπικό σιδηροδρομικό δίκτυο, περίπου 50 χιλιόμετρων. Το, σύστημα, το μεταφορικό σύστημα αυτό δεν επιβαρύνει καθόλου τις ε, οδικές αρτηρίες, αλλά μεταφέρει εμπορεύματα και συνδέει τους εσωτερικούς λιμένες με τους ε, σιδηροδρόμους. Τώρα, ε, το λιμάνι του Ντούσπουργκ έχει ε, διακινεί τεράστιο όγκο τόνους εμπαραβματοκιβωτίων. Όχι τόσους όσους το Ρότερνταμ φυσικά, αλλά αρκετούς. Και αυτός ο όγκος πρέπει να δούμε πώς θα μεταφερθεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Και αναφερθήκατε στις ε, γέφυρες που ανοίγουν και αυτές είναι κάτι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται η δημιουργία περισσότερων τέτοιων έργων υποδομής έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η διακίνηση των εμπορευμάτων. Τώρα αναφερθήκατε στο λιώσιμο των παγετώνων και αυτό είναι πράγματι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στάθμη του Ρήνου. Τα τελευταία χρόνια ήμασταν αρκετά τυχεροί με το θέμα αυτό, όμως είναι μια, ένας υπολογίσιμος ε, κίνδυνος. Και ανέφερε μάλιστα και το παράδειγμα της ε, BASF και του Ludwigshafen, που είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό παράδειγμα του πόσο αναγκαίες είναι οι κατάλληλες υποδομές. Διότι όταν μια τόσο μεγάλη εταιρεία όπως η BASF δεν μπορεί για δύο και περισσότερους μήνες να, ε, να λειτουργήσει εξαιτίας της στάθμης ε, του νερού και εξαιτίας των προβλημάτων σύνδεσης, είναι πάρα πολύ ε, είναι ενδεικτικό του μεγέθους του προβλήματος, του, της δικτύωσης των υποδομών. Στο Duisburg επενδύσαμε 200 εκατομμύρια ευρώ από τη δική μας τσέπη για τις διατροπικές ναι. υποδομές. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αναπτυχθεί και έχει αυξηθεί η χρήση μας ε, και η διακίνηση παραβηματοκιβωτίων. Χρειάζεται λοιπόν έργα και από εμάς. Κυρία Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να, να διευκρινίσω το θέμα της, ε, του εξυγχρονισμού στο έγγραφο σχετικά με το πρασίνισμα των σκαφών γίνεται, ε, αποδεικνύεται ότι όλα αυτά λειτουργούν πολύ, ε, μάλλον η εσωτερική λαυσιπλογία τα πάει πολύ καλά όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ωστόσο όχι τόσο καλά όσον αφορά τα οξύδια ζώτου και άλλους ρήπους. Οπότε εξετάζουμε τις ε, δυνατότητες εξυγχρονισμού των κινητήρων σε σχέση με αυτούς τους ρήπους. Παράλληλα, στον σιδηροδρομικό τομέα υπάρχει δυνατότητα ε, γιατί υπάρχουν χρήματα για να εξυγχρονιστούν ε, οι σύρμοι ως προς το θόρυβο. Και ενώ τα χρήματα για τα σκάφη ε, αφορούν τις εκπομπές ε, ρήπων στην ατμόσφαιρα. Τώρα όσον αφορά τα, τα, τους λιμένες εντός πόλεων, δεν χρειάζεται να πάει κανείς μακριά, υπάρχει το λιμάνι των Βρυξελών. Αν έχεις ας πούμε έναν οικοδομικό ε, οικοδομικές εργασίες ε, και έχεις ε, μπάζα να μεταφέρεις ε, πολύ καλά τα καταφέρνεις να περιορίσεις τον αριθμό των ε, φορτηγών, αν το κάνεις αυτό με φορτηγίδα ε, για μεταφορά δηλαδή των μπάζων στους ε, κατάλληλους χώρους. Το ίδιο γίνεται και με τα σούπερ μάρκετ που μπορούν να τροφοδοτηθούν μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών για σοβαριά πράγματα όπως τα ποτά για παράδειγμα. Α, ναι, και τα pub, και τα pub, τα μπαρ μπορούν να τροφοδοτηθούν έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ο Πέτερ και ο Δούναβης. Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση ήταν από την κυρία Μάισνερ. Σε ποια γλώσσα θα πρέπει να γίνει τρεις, τρεις ε, βασικές γλω... επίσημες γλώσσες. Γαλλικά, γερμανικά και ολλανδικά και γαλλικά, γερμανικά και ρωσικά. Και θα πρέπει να ξεχνάμε και τα αγγλικά. όχι επειδή μόνο ο πρόεδρός μας είναι Άγγλος, όχι, ε, είναι πολύ σημαντικό ε, θέμα η γλώσσα στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Η δεύτερη ερώτηση ήταν από τον κύριο Βαντάλεν σε σχέση με εκείνο το κομμάτι Φιλσκόφε δεν, έχουμε, δεν είχαμε ακόμα επαφή με το νέο κοινοβούλιο, τη νέα κυβέρνηση της κυρίας Μέρκελ, αλλά θα εστιάσουμε περισσότερο στον κάτω Δούναβη. Και ήδη είχαμε επαφές με του συναδέλφους της Γάμα Δέλτα Μούβ. αυτή θα πρέπει να το συζητήσουμε με την κυβέρνηση της Γερμανίας και εκείνο το κομμάτι, Open Στράουδινγκ, δεν είναι η μόνη συμφόρηση στο Δούναβη. Έχουμε και αλλού σημεία συμφόρηση. Στην Ουγγαρία 50 ε, Ρουμανία, Βουλγαρία. Επίσης έχουμε άλλο άλλη συμφόρηση, άλλα σημεία συμφόρηση. και άκουσα μάλιστα και κάποια πράγματα από την κυρία Τικάου για τον εξυγχρονισμό του στόλου. Νομίζω πω ο βασικός ρόλος ε, θα απεχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι όπως έχω πει εδώ και πέντε χρόνια δεν υπάρχει καμία εταιρεία ε, εφοπλιστική στο Δούναβι που να έχει κέρδη και μόνο ένα καινούριο σκάφο έχει φτιαχτεί. Μιλάμε για πρασίνισμα και νέε επενδύσει. Πώ μπορεί μια εταιρεία να βάλει λεφτά στο πρασίνισμα, αφού τσακώνεται και προσπαθεί, αγωνίζεται μάλλον για να επιζήσει. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Ξέρετε ότι είναι όλο χαμηλότερες ε, οι ε, επιβατικές ε, μεταφορές, ενώ στα φορτία όλο ένα και μειώνονται οι μεταφορές. Ε, ποιο θα βάλει λεφτά αφού δεν έχει λεφτά. Και την ερώτηση του πρόεδρου μας, του Μπράιεν, ρώτησε, είπε ότι ο Δούναβης δεν είναι πλωτός. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι πλωτός ο Δούναβης. Εγώ εργαζόμουν σε ένα επιβατικό πλοίο από το Ρότερνταμ στη Μαύρη Θάλασσα και Και αυτό το ονομάζαμε η γκρίζα ευρωπαϊκή περιπέτεια. Γιατί όχι λόγω του Ρήνου, αλλά λόγω του Δούναβη. Ο Δούναβη είναι πλωτό καθ' όλη τη διάρκεια του έτου. Από εμπορικό εκεί απόψεις όμως αυτό δεν αρκεί. Γιατί φέτος είχαμε και στο κοινό κομμάτι της Ρουμανίας Βουλγαρίας κοντά στην πόλη ε, της Βουλγαρίας είχαμε μόνο ένα 1,1 μέτρο. Ε, ένα μικρό παιδάκι, μπορείς να πας περπατώντας απέναντι. Ε, και αυτό είναι το βαθύτερο σημείο αυτό είναι πρόβλημα. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι αρχίζοντας από τη σκεπή. Πρέπει να ξεκινήσεις από τα θεμέλια. Και τα θεμέλια για το Δούναβι είναι υποδομή, αλλά για την ώρα υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης ορισμένων κρατών μελών. Αυτό και νομίζω ξεπέρασε το χρόνο μου. Ευχαριστώ επανέλθω στην ερώτηση της κυρίας Μάιστερ. Πώς να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τις ε, οδούς, τις εσωτερικές οδούς ναυσιπλοείας. Είναι θέμα κατάρτισης, πιστοποίησης, εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους ε, ε καπετάνιους των σκαφών κλπ. Και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Μισθή, η ημερομίσθια είναι πολύ χαμηλά για εκείνους που μπαίνουν ε, νεοφώτιστοι στον τομέα και αυτό σχετίζεται και με η κερδοφορία του τομέα. Αν δεν υπάρχει κέρδος δεν θα μπορεί κανείς να αυξήσει τους μισθούς ή τα ημερομίστια Όλο και πιο πολλοί άνθρωποι από την Ασία, από τις Φιλιππίνες εργάζονται στα σκάφη των εσωτερικών αυτών οδών. Και αν δεν αξίζει τον κόπο δεν θα έρθουν νέοι Ευρωπαίοι να εργαστούν στον τομέα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εφαρμογής συνέχειας. Μπορεί να ενδιαφέρεται κανείς να εργαστεί από τη στιγμή που θα μπορεί τελικά να γίνει κυβερνήτης του σκάφους. Αλλά ε, δεν υπάρχει δυνατότητα να αναρριχηθείς, δεν, σε προσελκύει. Είναι καλός ο τομέας για αυτούς που είναι περιπετιώδεις, αλλά μετά από 10 χρόνια πρέπει να φύγουν, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν στην καριέρα τους. Τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Να υπάρχει μια συνέχεια στην καριέρα κάποιου που μπαίνει στον τομέα. Πάνω από 50% των καπετάνιων είναι πάνω από 55. Άρα θα υπάρχει διαστοτικό πρόβλημα σε 10 χρόνια, αν δεν ανανεωθεί το προσωπικό. Λοιπόν, τι κάνει το ΣΕΦ, ήταν άλλη ερώτηση αυτή. 57% του τομέα είναι μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός. Αν ρωτάτε τι κάνει ο τομέας είναι δύσκολος. Οι εσωτερικές ε, οδύναυση πλοίας δεν μπορούν να επηρεάσουν τα σχέδια φόρτωσης, τις δραστηριότητε φόρτωσης. Οι μεγάλες εταιρείες ελέγχουν τους όγκους φόρτωσης, εκφόρτωσης. Άρα χρειάζεται βελτιστοποίηση της όλης αλυσίδας μεταφοράς των εμπορευμάτων. Αυτοί που χρησιμοποιούν, αυτοί που ελέγχουν, αυτοί που κυβερνούν τα πλοία, τα πλοία, δεν ελέγχουν τους ρυθμούς φορτοεκφόρτωσης. Και αν δεν ελέγχεις τα φορτία, εξαρτάσαι από τρίτα μέρη. Αυτά έχω να πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε το πρώτο τμήμα. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει ανάπτυξη τουρισμού. Διάφο... Μου έρχονται διάφορα φυλάδια για τις κουραζιέρες ε, την εταιρεία Viking ε, για κρουαζιέρες στα ποτάμια, άρα η πλευρά αυτή των επιβατών, των τουριστών ίσως ε, δώσει κάποια κέρδη και πόρους στα ποτάμια. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ όλους για τις ε, ομιλίες σας και τις απαντήσεις που δώσατε. Παρακαλώ, μπορείτε εσείς να αποχωρήσετε για να έρθουν οι επόμενοι τέσσερις προσκεκλημένοι. Κανένα λεπτό θα χρειαστούμε για την αλλαγή θέσεων, αλλά ευχαριστώ όλους σας που μιλήσατε. Ελάτε παιδιά, ελάτε παιδιά να συνεχίσουμε στην ώρα μας. Ήρθε ο κύριος Σίλιτο. Είναι εκπρόσωπος των Lloyds, του νεογνώμονα. Πάμε προς εξυγχρονισμένο στόλο των οδών εσωτερική ναυσιπλοεία. Κύριος Χάνς Βαντεβέρ ξεκινά. Η κυρία Χακστάινερ. Μετά ο κύριος Σίλιτο και ο κύριος Βαντεβέλ. Ο κύριος Βαντεβέρ, Γενικός Γραμματέας τη Κεντρικής Επιτροπής για την Αυσιπλοεία του Ρήνου. Μας αρέσει και ο Ρήνος. Εξίσου όπως και ο Δούναβης, κύριε Βαντεβέρ, σας το λέω αυτό, αλλά έχετε το λόγο και για έξι λεπτά τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως είμαι πολύ χαρούμενος που με καλέσατε. Είμαι τακτικός φιλοξενούμενος στην Επιτροπή σας και ήσασταν αρκετά, αρκετές φορές ήσασταν φιλοξενούμενος μας εσείς στο Στρασβούργο. Να πω κάτι για το CCNR η Επιτροπή μου θα παίξει βλέπετε βασικό ρόλο στην εκτέλεση του προγράμματος, στην υλοποίηση του προγράμματος Ναϊάδες. ε, χώρες του Ρήνου ε, συμμετέχουν σε αυτό το φορέα που ιδρύθηκε το 1815 και το 1868 η αποστολή καθορίστηκε ελευθερία και ευμάρεια όσον αφορά και δυνατότητα να ανθεί μάλλον η ναυσιπλοεία στο Ρήνο ήταν ο στόχος και τέθησαν πλαίσια για συνθήκες, για ισότιμες συνθήκες ε, για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αναφέρθηκε και πριν ότι όσον αφορά τη σημασία της εσωτερικής ναυσιπλοείας στην Ευρώπη μπορεί να πει κανείς ότι περίπου 60 με 70% της κυκλοφορίας στις εσωτερικές οδούς ναυσιπλοείας περνά από το Ρήνο. Έχουμε πέντε κράτη-μέλη, Βελγίο, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Ελβετία και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να πούμε εδώ ότι έχουμε στενή και αποτελεσματική ανοιχτή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φεύγουμε από το Ρήνο και κινούμαστε πιο πέρα από το ποτάμι, ρίχνουμε το βλέμμα μας και αλλού. Και ο φορέας μας καλύπτει όλο το σύστημα το μεταφορικό μέσο εσωτερικών οδών αυσιπλοίας στην Ευρώπη. Πρόσφατα ε, είχαμε ένα όραμα για το 2018, στόχους για το 2018, για να εναρμονίσουμε τις δραστηριότητες μας σωστά, εστιαζόμενοι επιβιωσίμου αναπτύξεως αυτού του τρόπου μεταφορών σε συντονισμό με τις πρωτοβουλίες του Ναϊάδες. Τώρα ασχολούμεθα με τα πλοία, με τα σκάφη σήμερα. Σχετικά με αυτό πρέπει να πω ότι ήταν, είναι εργαλείο των μεταφορών το πλοίο, αλλά είναι και αδυναμία του. Γιατί το λέω αυτό. Αργός ο ρυθμός του στόλου. Βλέπετε τα στοιχεία για τα υγρά φορτία, στεγνά φορτία και τις κουραζιέρες στα ποτάμια το μισό χρόνο τα, ο μισός τόλος είναι για, με σκάφη πάνω από μετά το 2000 στον τομέα των δεξαμενοπλοίων η παρόμοια κατάσταση αλλά όσον αφορά το ξηρό φορτίο είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, είναι παλιά τα πλοία και χαμηλή ρυθμή, ρυθμή Άρα έχουμε πολύ μακρύ κύκλο για την ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας. Άρα έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συντονιστούμε με τις πολιτικές προκλήσεις που εμφανίζονται. και να κινούμεθα με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον. Βλέπετε τι γίνεται με το στόλο σε σχέση με το χρόνο. Για τα διάφορα είδη φορτίων, υγρό φορτίο, ξηρό φορτίο, και έχουμε κύματα νεοτεύκτων πλοίων που δημιουργούνται αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή η ανανέωση δεν γίνεται με σταθερό ρυθμό και έχουμε ακμές στη γραφική παράσταση με υπερβολική, ε, υπερβολική δυνατότητα μεταφοράς και δημιουργούνται προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Η κατανομή των φορτίων εμπορευματοκιβώτια είναι μόνο 10% του συνολικού όγκου, το ξηρό φορτίο 2 τρίτα και 1 τέταρτο το υγρό φορτίο. Θυμηθείτε τα ποσοστά ανάπτυξης και τα νέα σκάφη όσον αφορά τα υγρά ε, φορτία. Βλέπετε πόσο σημαντικά είναι τα νέα σκάφη, τα νεότευτα σκάφη για τα δεξαμενόπλια, για τον τομέα των δεξαμενοπλίων. Πάμε στα, στο πρόγραμμα Ναϊάδες και την υλοποίηση του προγράμματος. Άρα, για να τα κάνουμε αυτά πρέπει να εξετάσουμε την περιβαλλοντική ποιότητα της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Πώς. Πρώτα απ' όλα, τυποποίηση της νέας τεχνολογίας. Χρειάζονται πλαίσια κατάλληλα για πιο γρήγορη ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας. Πρέπει να εφαρμόζονται όρια εκπομπών Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα των σκαφών να προσαρμόζονται στα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών ε, επιβλαβών αερίων και να λαμβάνουμε υπόψη και την οικονομική κρίση. Δεν χρειάζεται μόνο να προσαρμοστούν τα σκάφη στην νέα τεχνολογία. Χρειάζονται γενικέ υποδομέ. Η χρήση του υγροποιημένου αερίου, αερίου στην εσωτερική ναυσιοπλοεία απαιτεί συντονισμό για τις υπερκατασκευές των σκαφών. Και θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του τομέα. Ποιότητα διακυβέρνησης. Δύο λόγια, Πρόεδρε. Στενή συνεργασία μεταξύ του CNR και της DG Move στον τομέα των τεχνικών απαιτήσεων Τη της επαγγελματικής κατάρτισης και προσόντων του προσωπικού και στον τομέα της επίβλεψης της αγοράς. Πώς. Δυστυχώς δεν είναι ευανάγνωστες οι διαφάνειες. Με νέες δομές διακυβέρνησης. Οι οποίες εδράζονται επί της εμπειρίας της τελευταίας δεκαετίας. Μάθαμε πολλά. Και δείξαμε ότι μπορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του CNR και οι εμπορευόμενοι σε μια νέα δομή η οποία θα εξορθολογήσει τις ρυθμιστικές μας ελεγκτικές δραστηριότητε και θα δημιουργήσει μια βάση για ταχύτερη ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάντεβελτ η νέα Επιτροπή Μεταφορών ίσως ε, το φθινόπωρο θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτές ε, τις προτάσεις. Θα ήταν καλό λοιπόν ε, κάποια στιγμή στο Στρασβούργο να, καλέσει, να σας καλέσει η νέα Επιτροπή Μεταφορών. Έτσι μια ιδέα λέω. Η κυρία Τερίσα Χάκστα είναι η επόμενη Γενική Γραμματέας της EBU, της Ευρωπαϊκής <laughs> Ένωσης Εσωτερικής Ναυσιπλαιοίας και όχι της Eurovision. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή Μεταφορών που οργάνωσε αυτήν την ε, ακρόαση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ε, τομέα μας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εσωτερικής Ναυσιπλοείας. Είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών συνδέσμων ε, μεταφορέων που διαστηριοποιούνται στην εσωτερική ναυσιπλοεία στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ε, δραστηριοποιούνται στον ε, Δούναβη. Θα σας αναφέρω ορισμένα σημαντικά στοιχεία για ε, την εσωτερική ναυσιπλοεία. Η εσωτερική ναυσιπλοεία στην Ευρώπη μεταφέρει περίπου 500 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 130 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα χιλιομετρικούς τόνους είναι περίπου 5,6% της συνολικής μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ορισμένα κράτη-μέλη όμως το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο, όπως για παράδειγμα στις κάτω χώρες, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Χαρακτηριστικά τώρα της αστατονικής αναυσιπλοείας ε, είναι καταρχάς η μεγάλη οικονομία κλίμακας που έχει. Έχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από όλα τα μέσα μεταφοράς Χαρακτηρίζεται επίσης από ενεργειακή απόδοση και από απόδοση κόστους και από χαμηλό κόστος εξωτερικών δαπανών. Επίσης όμως χαρακτηρίζεται από το ότι λειτουργεί σε μια απόλυτα απελευθερωμένη αγορά και πραγματικά εξυπηρετεί πολύ μεγάλες αγορές και στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και των παραδοσιακών μεταφορών. Δεν ε, μεταφέρει όμως μόνο βαρύ φορτίο και εμπορευματοκιβώτια, όμως ε, και εξειδικευμένα εμπορεύματα σε συγκεκριμένες ε, περιοχές. Επίσης υψηλής σημασία έχει και η τουριστική κίνηση, η μεταφορά επιβατών, που όπως είπε και ο πρόεδρος, ε, άλλο και αυξάνεται, και επίσης οι αστικές ε, μεταφορές. Ένα επίσης χαρακτηριστικό του τομέα αυτού είναι η ε, καινοτομία που τον διακρίνει και η άμεση προσαρμογή στις νέες προκλήσεις. Τώρα θα σας αναφέρω τις ανάγκες του τομέα μας. Μια που μιλάμε για το πρόγραμμα ΝΑΙΑΔΕΣ 2, το οποίο υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πέραν αυτού όμως χρειαζόμαστε επίσης ισχυρές υποδομές και χρηματοδότηση από, την, από το Connecting Europe αλλά καθώς και από τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοείας μέσω των προτάσεων ε, στα πλαίσια του ΝΑΙΑΔΕΣ 2, για παράδειγμα στον τομέα της μετάσκευή και εξυγχρονισμού των πλοίων, αλλά και προγραμμάτων τα οποία θα ε, είναι διαθέσιμα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Τώρα, όσον αφορά συγκεκριμένα το πρόγραμμα ΝΑΙΑΔΕΣ, σημαντικό είναι η ποιότητα της υποδομής, η καινοτομία του στόλου και σε αυτό θα επανέλθω πολύ σύντομα, η ομαλή λειτουργία του αγοράς, ε, το καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και οι ε, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Πρωτού αναφερθώ όμω στην καινοτομία που είναι το κυριότερο σημείο, να σας ε, υπενθυμίσω κάτι που έχει συζητηθεί στο προηγούμενο πάνελ, την ποιοτική υποδομή δηλαδή, η οποία από την άποψη του χρήστη είναι, ε, είναι απαραίτητη προϋπόθεση διότι χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει εσωτερική ναυσιπλοεία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχουμε πάνω από 36.000 χιλιόμετρα εσωτερικών πλωτών οδών και εκατοντάδε εσωτερικούς λιμένες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορούν να απορροφήσουν έναν πολύ μεγαλύτερο όγκο κίνηση και μεταφορών και να ε, μειώσουν το πρόβλημα της συμφόρησης. Τώρα, επανέρχομαι στο θέμα της ε, καινοτομίας. Όπως σας είπα, υπάρχει τεράστιο δυναμικό στον τομέα αυτό. Είναι ενεργειακά αποδοτικός, οικονομικά αποδοτικός. Χρειάζεται βέβαια πρασίνισμα του στόλου, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις του προγράμματος Εναϊάδες μέσω της μετασκευής των πλοίων, αλλά και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Και εδώ να αναφερθώ και να υπενθυμίσω ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι για εμάς ε, ένα πολύ υποσχόμενο καύσιμο για τα νέα σκάφη και εμείς ε, παροτρύνουμε την ε, χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου στα σκάφη ως αναλλακτική πηγή καυσίμων. Αυτό βέβαια χρειάζεται και κατάλληλη νομοθεσία. Εδώ έχετε, βλέπετε ορισμένα παραδείγματα των πρώτων σκαφών τα οποία ε, πλέον τι εσωτερικέ επιλωτές οδούς με αυτό το ευρωπημένο φυσικό αέριο εδώ και ένα-δύο χρόνια. Τώρα, ε, μιλώντας για καινοτομία και καινοτομία στο στόλο, εδώ να, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ορισμένες ε, προτάσεις έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στο στόλο να εξυγχρονιστεί και να ανακαινιστεί. Επίσης υπάρχει μια τεχνικής φύσης οδηγία η οποία προτείνει τίνει νέα εναρμονισμένα πρότυπα που θα ισχύουν πανευρωπαϊκά έτσι ώστε να ε, χρησιμοποιηθούν τα, πρότυπα, τα υψηλά πρότυπα του ρήνου σε όλη την Ευρώπη και η δεύτερη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια τροποποίηση της υφιστάμεν, του φυστάμενου κανονισμού για την χωρητικότητα του στόλου. Αυτό, αυτή η πρόταση θα στήσει δυνατό να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή και να χρησιμοποιηθούν τα ε, αποθεματικά ταμεία για το πρασίνισμα για παράδειγμα. Και σε αυτό το σημείο ζητούμε από το Κοινοβούλιο να στηρίξει την πρόταση αυτή. Ολοκληρώνοντας τώρα, τι σημαίνει το πρόγραμμα Αναϊάνδες 2 για τον ε, κλάδο μας. Θα θέλαμε καταρχάς να πούμε ότι πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα Ναϊάδες μαζί με τα υπόλοιπα ε, ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να ενσωματωθούν στους ε, στόχους και να υλοποιήσουν τους στόχους της βελτίωσης των εσωτερικών ε, ε, πλωτών μεταφορών. Όμως χρειάζεται και η διασφάλιση χρηματοδότησης πέρα από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Και σε αυτό το σημείο κάνουμε έκκληση στο Κοινοβούλιο να στηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να στηρίξει τη βιομηχανία με το να καταστήσει δυνατή αυτή τη νέα πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριος Άντριου Σίλιτεο στη συνέχεια θα μας παρουσιάσει την ε, εκτίμηση κινδύνου που έχει κάνει η εταιρεία Lloyds. Lloyds Register Marine. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να εστιάσω στην ε, καινοτομία, ιδιαίτερα στο Στόλοφ και θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα του πώς αυτό έχει πραγματοποιηθεί σε ε, σκάφη αλλά και σε μελλοντικά προγράμματα. Καταρχάς, να πω ότι οι εσωτερικές πλωτές οδοί μας δίνουν μια καλή ευκαιρία για ε, καθαρή και ε, βιώσιμη ε, ναυσιπλοεία και βιώσιμε μεταφορές. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο η βιομηχανία θα κάνει να βγούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά, η κοινωνία των πολιτών αλλά και οι οικονομικοί παράγοντες έχουν πολύ μεγάλο συμφέρον για, ε, για αυτό. Η μείωση κόστους, μείωση χρήσης καυσίμων και η χρήση υγροπημένου φυσικού αερίου θα βοηθήσει σε αυτό. Το πακέτο Ναϊάδες 2 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα εναλλακτικά καύσιμα, ιδιαίτερα στο υγροποιημένο φυσικό αέριο και αυτή είναι μια τεχνολογία την οποία βλέπουμε να χρησιμοποιείται με επιτυχία τον τελευταίο καιρό. Επίσης, ε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η κίνηση με βιοντίζελ, διότι πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα ελέγχεται καλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Τώρα, για τα σκάφη των εσωτερικών ε, πλωτονοδών, οι ενεργειακές και ανάγκες ε, διαφέρουν πάρα πολύ ανάλογα με το αν ανεβαίνουν ή αν κατεβαίνουν έναν ποταμό. Η χρήση επίσης του υδρογόνου είναι μια πολύ καλή πιθανή λύση, καθώς και η κατασκευή ελαφρύτερων πλοίων. Λοιπόν, χρειάζονται κατάλληλες υποδομές που θα έχουν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη χρήση αυτής της επιλογής. Το υγροποιημένο αέριο είναι μια επιλογή και τα πρώτα σκάφη ήδη ε, είναι σε υπηρεσία Βλέπετε ένα τάνκερ που χρησιμοποιεί και τα δύο είδη καυσίμων, υβριδικό και είναι το πρώτο από τα σκάφη που χρησιμοποιεί το υγρό. Βλέπετε το Green Stream προϊόντα σε χημικά τάνκερ που χρησιμοποιούν σαν καύσιμο το υγροποιημένο αέριο. Είναι ένα νέο καύσιμο για τα σκάφη για την εσωτερική ναυσιπλοεία και οι κανονισμοί είναι πίσω από την τεχνολογία. Άρα η πιστοποίηση πρέπει να βασίζεται επί παρεκκλήσεων μετά από ένα σχεδια... διαδικασία σχεδιασμού και έγκρισης που βασίζεται στην ανάλυση του κινδύνου. Θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα για να, να επιτρέψουμε στους κανόνες να χρησιμοποιείτε το υγροποιημένο αέριο. Να δώσω και άλλα παραδείγματα για να σας δείξουμε ότι είναι, πρακτική, είναι πραγματικότητα ο σύγχρονος στόλος και δεν είναι απλώς κάτι θεωρητικό. Παραδείγματα βλέπετε τα tanker I, τύπου I που χρησιμοποιούν το υγροποιημένο αέριο σαν καύσιμο και βλέπετε την, ε, το σκάφος ε, που προωθεί τις ε, σπρώχνει κινή, κινή τις φορτηγίδες που χρησιμοποιεί ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτού του είδους το καύσιμο με αλλαγή τροποποίηση. Το Άγγερ έγινε ε, δύο είδη καυσίμων και το Ευρωπαϊκό Περίπου ε, χρησιμοποιεί ε, χώρο βέβαια το κύλινδρος για να μπει το αέριο παίρνει, αφαιρεί κάποιο, κάποια δυνατότητα μεταφοράς φορτίου αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη, μεγάλο ποσοστό μπορούμε στο σχεδιασμό ενός σκάφους να λάβουμε υπόψη τη χρήση νέου καυσίμου και μπορούν να γίνουν ε, μετασκευές των σκαφών σε κάποια φάση της ζωής τους όπως αντικατάσταση του κινητήρα. Γενικά αυτό όμως τελικά θα αποσβεστεί μέσω των κερδών ε, με την αύξηση των ορών ε, που πλέει το πλοίο. Και έχουμε μετά το δεξαμενόπλιο Άργος βλέπετε ερευνούμε την έννοια και θέλουμε ε, να μεταφέρει το, ε, το υγροποιημένο αέριο. Δεν, δεν μπορεί να μεταφέρει κανονικά, δεν μπορεί να μεταφέρει το υγροποιημένο αέριο σαν φορτίο στην εσωτερική πλοή και θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες για να επιτρέπεται. Για το τάνκερ μεταφοράς αερίου ερευνούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε δει ταυτόσιμα πλοία που παράγονται που θα μπορούν να χρησιμοποιούν δύο είδη καυσίμων. Έχουμε και άλλα προγράμματα τα οποία επεξεργαζόμαστε, σε αρχικό σχεδιασμό βρισκόμαστε για να δώσουμε μια γεύση σχετικά με το οποίο θεωρείται σαν τεχνικά εφικτό βλέπουμε ε, μεταφο σκάφος μεταφοράς ε, ξηρού καυσίμου ε, και δύο ε, δεξαμενόπια και μετά δύο, ηλεκτρικά, ε, δύο σκάφη που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια και υγροποιημένο αέριο και είναι οχηματαγωγά και ένα άλλο είδος οχηματαγωγού σας έδειξα λοιπόν ότι τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοείας δίνουν δυνατότητες για να αναπτύξουμε ένα πιο σύγχρονο στόλο μέσω νέας τεχνολογίας. Υπάρχει καινοτομία εντός του τομέα αυτού αλλά δεν είναι κάτι που είναι και μοναδικό, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Υπάρχει τεχνολογία, έχουν γίνει έρευνε έρευνες, η τεχνολογία για τα μεγάλα σκάφη ανοιχτής θάλασσας τα ποντοπόρα πλοία και οι νιογνώμονες ε, συμμετέχουν στην ε, όλη προσπάθεια και μπορούν την εμπειρία τους να τη δώσουν φάση τεχνικές επιδόσεις και τα θέματα ασφαλείας. Να συμμετάσχουν οι νιογνώμονες. Εναλλακτικά καύσιμα και κυρίως το υγροποιημένο φυσικό αέριο έχουν αποδείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν αλλού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα και για τα σκάφη εσωτερική αυτοπλοεία. Είναι καλύτερο αυτό να το, να το εντάξουμε σε ένα νέο σκάφο, σχεδιασμό νέου σκάφου, αλλά μπορούμε να μετασκευάσουμε και φυστάμενα ε, σκάφη σε κάποια φάση τη ζωή του σκάφου να γίνει κατάλληλη μετασκευή, να χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο. Ευχαριστώ πολύ, Άντριου. Επόμενο Χάνκ Βαντεβέλτ τώρα που είναι Γενικό Γραμματέα ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, Πλειοκτητών. Σας ευχαριστώ. Ε, ναι. ε, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνητών, Καπετάνιων. Με συγχωρείτε. ο, ο οργανισμός μας ασχολείται με τα συμφέροντα των καπετάνιων και άκουσα κάποιες ε, αρνητικά σχόλια σε σχέση με τους ε, οργανισμούς ότι ακολουθούν ε, κάποιες οικογενειακές δομές και ότι αναδιοργανώ... εγώ πιστεύω πως κάνουμε πολύ καλή δουλειά, αναδιοργανώνουμε τα πράγματα και γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ευρωπαϊκό το πρόγραμμα Ναϊάδας και το πρώτο και το δεύτερο. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο έχουν κάνει καλή δουλειά, αλλά πρέπει να υπάρξει ισορροπία εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία βεβαίως, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ε, σε ένα ισότιμο πεδίο για όλους και με πλήρη ενημέρωση προς όλους. Ε, η αγορά των εσωτερικών πλωτών οδών υποφέρει από έλλειψη ισορροπίας εδώ και πέντε χρόνια και αυτό οδηγεί στην ε, διατάραξη της αγοράς. Βλέπουμε ότι η χωρητικότητα των στόλου περνάει κρίση, ε, τα σκάφη πρέπει να είναι όλο ένα και πιο ειδικευμένα και άρα ε, αυτό συνεπάει, ε, μάλλον έχουμε δει ταυτόχρονα και μείωση της ζήτησης όσον αφορά την βιομηχανία, την μεταλλουργία αλλά και τη, τον κλάδο των οικοδομών, τον κατασκευαστικό και Βλέπουμε ένα σωρό πράγματα που γίνονται, επηρεάζουν την νομοθεσία, χωρίς όμως να αλλάζουν τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Τώρα, επίσης είδαμε τα σκάφη διπλού και κήτους ε, να αναπτύσσονται και υπερβολική χωρητικότητα στα μεγάλα πλοία δεν επηρεάζει τα, μικρά, γιατί υπάρχει ανταγωνιστικότητα ανάμεσά τους και χάνουν και τα μικρότερα φορτία. Και τελικά αυτό οδηγεί σε καταστροφική κατάσταση, διότι λείπουν οι επενδύσεις, αλλά υπάρχει και το θέμα της ε, ελκυστικότητας του τομέα για επενδυτές. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αγορά αυτή τη στιγμή είναι βέβαιη και αυτό είναι και πολύ αρνητικό. Ε, ε, είμαστε, έχουν εξαντληθεί τα ενεργητικά, αυτή τη στιγμή καταναλώνουν τα αποθυματικά και μάλιστα κάποιες εταιρείες βυθίστηκαν. Ε, ε, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να μην προσπαθούμε με τα ίδια μέσα να συνεχίσουμε. Υπάρχουν πολλές εθνικές ομοθεσίε που λειτουργούν κατά της εισόδου ξένων αλλοδαπών. Αυτό δεν βελτιώνει τον ανταγωνισμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε ε, ε, ακόμα και ξένες εταιρείε. Ίσως αυτό να είναι υπερβολικό, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Ε, εάν δεν μειωθεί χωρίς μάλλον να μειωθεί η ανεξαρτησία των ε, επιχειρήσεων. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της διπλής, της μεγάλης χωρητικότητας, αλλά και τα τέλη, το κόστος κατασκευής νέων σκαφών ε, ε, ε, υπάρχουν και τα ναύλα τα οποία πρέπει να καθορίζονται με σωστό τρόπο. Εν τω μεταξύ η οικοδόμηση ενός νέου σκάφους παίρνει τουλάχιστον δύο χρόνια. πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη και πρέπει να προσθέσουμε εδώ και τις, κατασκευ... τις, τις παραγγελίες για την οικοδόμηση νέων σκαφών. Ένα δεύτερο θέμα που έχουμε είναι το μόνιμο μέσο χειρισμού της χωρητικότητας που είχαμε πριν από 10 χρόνια και λειτουργήσε πολύ καλά. Ε, και επίσης η ε, χορήγηση πιστώσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι πρόβλημα. Ε, πριν την οικονομική κατάρρευση πολλά χρήματα δίνονταν και γι' αυτό καταλήξαμε στην τρέχουσα υπερχωρητικότητα. Τώρα όμως ούτε με το σταγονόμετρο δεν βλέπουμε να δίνονται χρήματα ούτε καν για νέους κινητήρες για παράδειγμα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους καπετάνιους και τους ε, μεταφορείς για να δουλέψουμε επίση όρει, έτσι ώστε να φτιάξουμε μια πολύ στεναρή αλυσίδα, να δουλέψουμε στην διατροπικότητα, ε, να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τα πράγματα, να δημιουργηθεί υγιής ανταγωνισμός, ε, να βελτιώσουμε δηλαδή την επιμελητή αλλά και την οικονομική οικονομική πτυχή ε, του κλάδου. Να μιλήσω και για το άρθρο 8 που αναφέρθηκε ε, όσον αφορά τον κανονισμό του 99, η συγκήτρια στην χρωματότησή της μιλά για την αλλαγή του άρθρου 8. Αλλά πραγματικά υπερβάλλει, γιατί... Ε, το άρθρο 8 είναι ένα απόσπαστο τμήμα της ε, νομοθεσίας. Η εκτέλεση θα πρέπει να γίνεται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ε, του κλάδου κάθε φορά. Δεν μπορεί να ε, το ζητά μόνο όποτε το επιθυμεί. Γι' αυτό και ζητώ από την εισηγήτρια να αποσύρει τις σχετικές τροπολογίες. Νομίζω πως ε, θα πρέπει να μιλήσουμε και για την διατροπικότητα. Χρειάζεται να χειριστούμε τις κοινωνικές και τεχνικές πτυχές και πιστεύω πως ε, τα υπόλοιπα θα ρυθμιστούν. Είμαστε ευτυχεί δεν που μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σε αυτό το θέμα. Κυρία Μάισνερ, ε, τώρα, και θέλω να είστε σύντομοι παρακαλώ για να μείνουμε μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχουμε προκαθορίσει. Μάισνερ Βαρντάλ Κούν για την ώρα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καταρχάς, ε, μια ερώτηση στο και στον κύριο Βαντερβέρφτε όσον αφορά το όραμά σας για το 2018. Ε, κοίταξα την παρουσίασή σας και έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, ε, θέλετε να, ο τομέας να ενισχύσει την δική του ευθύνη και να ενισχυθούν οι προδιαγραφές. Αυτό για τους φιλελεύθερους φυσικά ακούγεται μελωδικό, μελωδικότατο. Όμως πρέπει να δούμε και πώς αυτό θα υλοποιηθεί. Και αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Έπειτα, όσον αφορά τις γλωσσικές ε, απαιτήσει που ε, αναφέρεται στο όραμα για το 2018, θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η γλώσσα θα είναι τα αγγλικά ή αν όχι ποια άλλη. Κυρία Χακστάινερ, καταρχάς, ήδη το αναφέρατε, όμως θα το ξαναρωτήσω. Αναφέρατε λοιπόν για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τη δυνατότητά τους να αναλάβουν πολύ μεγαλύτερο όγκο κίνηση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Μας αναφέρατε ε, το πρόβλημα του Δούναβη και την κατάσταση ε, στο Ρήνο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι χρειάζεται, τι είναι αναγκαίο έτσι ώστε να υλοποιηθούν τα προγράμματα αυτά και αν έχετε κάποια συγκεκριμένα νούμερα και συγκεκριμένους αριθμούς του πόσο θα κοστίσει αυτό. Τώρα, στον κύριο Σίλιτοου. Ε, αναφερθήκατε στο πρασίνισμα και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ την δυνατότητα χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου. Γι' αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ε, τι προβλέπετε, αν προβλέπετε κάτι τέτοιο ε, στην έκθεση, αν προβλέπετε κάποια μετασκευή των ε, ποτάμιων πλοίων έτσι ώστε αυτά να λειτουργούν με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Υπάρχουν επενδύσεις και τι σημαίνει αυτό για τους επλειοκτήτες. Τώρα, Αναφερθήκατε στην ε, ανασφάλεια που επικρατεί στις αγορές, στην ανασφάλεια στη... όσον αφορά τις ε, πιστώσεις. Εδώ θέλω, θέλω να ρωτήσω αν τα αποθεματικά ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τι μπορεί να γίνει επιπροσθέτω. Ε, αναφερθήκατε ήδη στη διαφάνεια της αγοράς, ε, στις πρώτες για το 2018. Τι ακόμα μπορείτε να φανταστείτε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πέτερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η πρώτη μου ερώτηση είναι προς την κυρία Χακστάινερ και στον κύριο Φοντερβέλτ για το νέο άρθρο 8. το οποίο ανέφεραν και αρκετοί προλαλήσαντες. Στο νέο λοιπόν άρθρο 8 αναφέρονται πράγματα όπως για παράδειγμα ανεξάρτητα από ό,τι αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, το οποίο είναι το βασικό, χρειάζεται ομοφωνία και ομόφωνη συμφωνία έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν τα ταμεία. Ο τομέας ποτέ δεν ε, χαρακτηρίστηκε από ομοφωνία και αυτό ισχύει και στην περίπτωση των αποθεματικών ταμείων. Εντάξει, όσον αφορά την οικονομία της Γερμανίας και της Ολλανδίας, τα αποθεματικά ταμεία είναι φραγοδίφρακα κανονικά. Όμως αυτό δεν ισχύει για όλους. Πώς λοιπόν μπορούμε να αγγιηθούμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον και θα υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες που έλειπαν. Έπειτα, κύριε Χακστάινερ, Κανείς δεν κατάφερε να με πείσει να υπερψηφίσω την πρόταση αυτή, θα ήθελα να σας πω. Και τι εννοώ με αυτό, ότι το νέο άρθρο 8 για την ε, πρόταση σχετικά με τη χωρητικότητα πιστεύω, αν το κατάλαβα καλά, ότι μας δίνει ένα πλεονέκτημα επιπλέον και αυτό είναι ότι οι καπετάνιοι θα μπορέσουν να έχουν ευκολότερη χρηματοδότηση ευκολότερη πρόσβαση στις ε, πιστώσεις για νέα πιο φιλικά προς το περιβάλλον σκάφη. Όμως, αυτό είναι το μοναδικό πλεονέκτημα που μπορώ να βρω από όλη την πρόταση. Και δεν νομίζω πως αυτό είναι κάτι που μπορούμε να δεχτούμε. Όπως είπε και ήδη ο κύριος Εφαντερφέλτ, υπάρχουν ορισμένοι κυβερνητές οι οποίοι δεν ε, βγάζουν αρκετά χρήματα για να ζήσουν, πόσο μάλλον αρκετά χρήματα για να επενδύσουν σε νέες μηχανές και σε νέους κινητήρες. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Ποιος λοιπόν μπορεί να μου εξηγήσει, ε, να με πείσει να ψηφίσω υπέρ αυτής της πρότασης. Αυτή η πρόταση δεν φαίνεται να αλλάζει απολύτως τίποτα για τους ε, καπετάνιους. Δεν φαίνεται να τους βγάζει από τη μιζέρια στην οποία ζουν σήμερα. Ο κύριος Κούν, ευχαριστώ πολύ για τις εισηγήσεις σας. Να σας ευχηθώ και καλή χρονιά όλας. Και το καλή χρονιά και να πάνε όλα καλά σημαίνει επίσης ότι εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στις εσωτερικές επιλωτές οδούς και στην αποφυγή όσο το δυνατόν περισσότερων ατυχημάτων εκεί. Και αυτό συνδέεται και με την ερώτηση που έχω προς τον κύριο Βαντερβέρτ και την κυρία Χακστάινερ, τον κύριο Σίλιτο και την κυρία Φαλεφέρτε, σε όλους σας δηλαδή. Τι γίνεται με τα πρότυπα ασφαλείας για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Πώς αυτά θα εφαρμοστούν και θα εξισορροπηθούν στο μέλλον. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, μεταφορά φορτίων στο Δούναβι, πώς θα, μπορούν θα αποφευθούν οι συγκρούσεις και μας ε, παρουσιάσατε κύριε Σίλητο ότι χρειάζονται καλύτεροι κινητήρες, νεότεροι, πιο φιλικοί προς το περιβάλλον όμως όσον αφορά την αποφυγή των συγκρούσεων υπάρχει κάποια νέα πρόοδος στην έρευνα, χρειάζεται κατάρτιση, νέα κατάρτιση των πληρωμάτων έτσι ώστε να μπορούν αυτά να χειριστούν τα νέα αυτά συστήματα που θα έχουν στη διάθεσή τους. Τέλος, στο προηγούμενο πάνελ συζητήσαμε για την ε, υποδομή και πώς θα την βελτιώσουμε έτσι ώστε να, να αποφύγουμε τις ε, συμφορήσεις. Αναφερθήκαμε στους ε, ναυπηγούς και θα ήθελα λοιπόν εγώ να σας ρωτήσω εσείς πώς θεωρείτε ότι μπορούν να προσαρμοστούν τα νέα αυτά πλοία στις ε, συνθήκες των ποταμών. Ας μην μιλάμε μόνο για την υποδομή στα λιμάνια, αλλά και στα νέα μοντέλα πλοίων τα οποία θα είναι πιο αποδοτικά και θα μπορούν να προσαρμοστούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια ερώτηση εγώ για τον κύριο Σίλιτο και αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δέχομαι τα εναλλακτικά καύσιμα και είναι βασικό τέτοιο καύσιμο το LNG. Αν δείτε την έκθεση του κύριου Φινάνσες που ανέφερε η κυρία Μάισνερ Υπάρχουν και άλλα στοιχεία εναλλακτικών καυσίμων που εμπεριέχονται. Η εθανόλη, παραδείγματο χάρη. Και αν δείτε τι κάνει ο Σταν ε, με, το, με την εθανόλη. Αλλά νομίζω ότι είναι σαν ένα καλάθιλο τα αυγά της του εναλλακτικού καυσίμου, δηλαδή στο LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και εγώ ανησυχώ λίγο γι' αυτό. Γιατί το λέω. Τέτοιου είδους πολιτικής δεν είναι σωστή. Και είναι και το θέμα της αποθεματοποίησης, της φύλαξης του υγροποιημένου αέριου. Δεν είναι εύκολο να αποθηκευτεί σε μείον κάποιους βαθμούς Κελσίου. Χρειάζεται κατάλληλη υποδομή και αυτό είναι ένα από τα ωφέλη χρυσέως της εθανόλης αντί του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και γιατί προβληματίζομαι. Έχουμε τη Στέρνερ που είναι πλειοκτήτρια εταιρεία που χρησιμοποιεί την εθανόλη. Κάποιος άλλος ακολουθεί το φυσικό αέριο, κάποια άλλη εταιρεία. Και ανησυχώ μήπως τελικά καταλήξουμε σε μια κατακαιρματισμένη προσέγγιση. Εσείς λέγατε όμως φυσικό αέριο, φυσικό αέριο, φυσικό αέριο συνέχεια. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ, εξετάστηκαν για την εσωτερική ναυσιπλοεία όπως η εθανόλη, παραδείγματος χάρη. Για τρία λεπτά με τη σειρά. Ο κύριος Βάντερ Βερμπ, Ξεκινά ο Χάντς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που ρώτησε η κυρία Μάισνερ. Το να συμπεριλάβουμε τη διαχείριση των πλειοκτητριών εταιριών στα θέματα ασφαλείας, αυτό το κάναμε για να αποφύγουμε λεπτομερές τεχνικές προδιαγραφές και για να χρησιμοποιήσουμε τη φιλοσοφία και τις ικανότητες των εταιριών για να καταφέρουμε να έχουμε κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας. Σε άλλους κλάδους έχουμε διαφορετικά παραδείγματα το πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να ακολουθήσουμε την ίδια προσέγγιση και για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Όσον αφορά τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις μεταφορές εσωτερικής ναυσιπλοείας, έχουμε προχωρήσει. Έχουμε σχέδιο συστήματος ορολογίας για τον τομέα. Βραχυπρόθεσμα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ξεπεράσουμε τους φυστάμενους κανόνες. Δηλαδή, στο Ρήνο είναι τα γερμανικά που χρησιμοποιούνται και η γλώσσα των παροχθείων χωρών χρησιμοποιούμε παρόμοιο σύστημα με τη ρωσική και γερμανική γλώσσα. Μαζί με την ορολογία και το έγγραφο, με την ορολογία της ποτάμιας ναυσιπλοείας, river speak στα αγγλικά, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Αυτά. Ως απάντηση στην ερώτηση που μου απευθύνθηκε προσωπικά. Ευχαριστώ, η κυρία Χακστάινερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη που έθεσαν ερωτήσεις. Καταρχάς, η ερώτηση που αφορά τη διαθεσιμότητα χώρου στα ποτάμια. Μάθαμε ότι στο Ρήνο υπάρχει δυναμικό που δεν χρησιμοποιείται. Μπορούμε να διπλασιάσουμε τον όγκο που μεταφέρει το Ρήνο. Στο Δούναβι ίσως έχουμε, μπορούμε να έχουμε 20 πλάσια, 20 όγκο. Αλλά πρέπει να υπάρχουν σωστοί όροι που εφαρμόζονται, σωστή στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη οικολογικές απαιτήσεις, οικονομικές. Και η στρατηγική για το Δούναβι παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το τομέα. Πιστεύουμε όμως ότι σύντομα η ανάπτυξη εφαρμογή των σχεδίων για τους διαδρόμους θα, παίξουν σημαντικό ρόλο, θα παίξει σημαντικό ρόλο. Χρειάζεται σωστή δίκαιη ισορροπία για να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό που υπάρχει. Τη χωρητικότητα. Το άρθρο 8, η τροποποίηση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χωρητικότητα του στόλου. Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό να επεκτείνουμε τη χρήση του πλαισίου αυτού, να χρησιμοποιήσουμε κοινωνικές πτυχές. Να μειώσουμε το βάρος που τίθεται στην αγορά. Θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο του Ναϊάδες και την γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική έτσι μεταφορές. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το αποθεματικό ταμείο και για μέτρα πρασινίσματος συνεργαζόμαστε όλοι αρμόδιοι και μπορούμε να πετύχουμε μια κοινή θέση για τη χρήση του Ταμείου. Θα ήταν επωφελές για όλους. Χρειαζόμαστε πρασίνισμα των σκαφών. Όμως περνάει μεγάλη κρίση για την ώρα ο τομέας. Ελπίζουμε να ανακάμψει τα επόμενα έτη. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα για αυτές τις απαιτήσει. Και γι' αυτό σας απευθύνω έκκληση να υποστηρίξετε τις προτινόμενες τροπολογίες. Τέλος, τα θέματα ασφαλείας που έθιξε ο κύριος Κούν. Η ασφάλεια είναι σοβαρότατο κριτήριο για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Έχουμε τις ψηλότερες προδιαγραφές όσον αφορά για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. Υπάρχουν διεθνείς προδιαγραφές που έχουν ναι, εξεταστεί και έχουν θεσπιστεί στη Γενέβη. Οι πλειοκτοί επιβάλλονται, οι πλειοκτήτες ξεπερνούν και τα όρια ασφαλείας. Ήψιστες οι προδιαγραφές για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. Ε, έχουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές στην Ευρώπη και ίσως όλο τον ε, κόσμο. Ευχαριστώ κύριο Σύλλητο. Ευχαριστώ. Ερώτηση της κυρίας Μάισνερ πρώτα απ' όλα. Για το υγροποιημένο αέριο σαν καύσιμο και τις υποδομές. Είναι αν το αυγό έκανε την κότα, η κότα το αυγό. Το χρησιμοποιούν το προϊόν αν υπάρχει και ερωτηματικό όσον αφορά το κόστος του φυσικού αερίου σαν καύσιμο. Οι αποφασίσεις για επενδύσεις ε, εξαρτώνται από την εξέταση των προγραμμάτων από τα ποντοπόρα πλοία. Αν βλέπουμε ότι όταν υπάρχει υποδομές, ο κόσμος ενδιαφέρεται. Η επένδυση στις υποδομές βελτιώνει την χρήση και απορρόφηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος, ενός καυσίμου. ως Βαντάλεν, ποια ωφέλη βλέπουμε. Βελτιώνει νέα τεχνολογία που θα χρησιμοποιείτε, μάλλον θα καλείτε τους κανονισμούς, δυνατότητα χρήσεως αναλλακτικών καυσίμων να χρησιμοποιείτε το υγροποιημένο φυσικό αέριο και σαν φορτίο. Να προχωρήσουν οι κανονισμοί για να συντονιστούν με την τεχνολογία που εξελίσσεται. Πολύ συχνά μένουν πίσω οι νόμοι από την τεχνολογία και χρειάζεται προσπάθεια συντονισμού. Αλλά όταν υπάρχει δυνατότητα συντονισμού Νομοθεσία με την τεχνολογία, αυτό είναι πάντα κάτι χρήσιμο να γίνεται. Ερώτηση του κ. Κον. Ναι. Αποφυγή συγκρούσεων είναι ύψιστη προτεραιότητα. Όλη η έρευνα και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται έχει αυτό το στόχο. Και η, και η χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου και η μεταφορά φυσικού υγροποιημένου αερίου ε, συνεπάγεται αποφυγή συγκρούσεων και πώς να αποφύγουμε τα αρνητικά αποτελέσματα αν υπάρξει ε, σύγκρουση, να είναι πιο ισχυρές οι δεξαμενές κλπ. Πιο ενισχυμένες. Βέβαια, ε, όπως όποτε φοράει κανείς τη ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο, φορά τη ζώνη ασφαλείας μήπως χρειαστεί, αλλά δεν θέλει να συγκρουστεί. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε, αποφύγουμε τις συγκρούσεις, αλλά κάνουμε και ό,τι χρειάζεται, παίρνουμε μέτρα ασφαλείας και ενισχύουμε τα σκάφη, αν ε, συμβεί μια σύγκρουση και μεταφέρουμε τελικά και από άλλες εμπειρίες μας ε, από τα ποντοπόρα πλοία, εμπειρίες στα, στα πλοία των ποταμών στον πρόεδρο ε, ε, συγκεντρωθήκαμε όσον αφορά στο φυσικό αέριο γιατί έχουμε μεγάλη εμπειρία, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το φυσικό αέριο μαθαίνουμε μαθήματα, υπάρχει ενδιαφέρον χρήσεως αυτού, υπάρχουν εναλλακτικέ, όπως είπατε, εθανόλοι, ε, κυψέλες καυσίμων, ηλεκτρική ενέργεια Αντί να παράγονται από του κινητήρε, να παράγεται ο, ο, ηλεκτρισμό από του κινητήρες όταν πλέει το σκάφος και παράγει ε, ε, ρήπου, να φορτίζονται μπαταρίες πιο πριν. Θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους εκπομπών διεξουδίου του άνθρακο, ε, αζωτούχων κλπ. Το αγροποιημένο λοιπόν φυσικό αέριο είναι μία λύση, όχι μόνη λύση. Ευχαριστώ ο κύριος Βαντεβέλτ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Διάφορες ερωτήσεις μου ετέθησαν να προσπαθήσω να συνοψίσω. Η κυρία Μάισνερ αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές. Κανείς δεν θέλει να επενδύσει. Δεν μπορεί να επενδύσει, διότι δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει η περίοδος αβεβαιότητας. Το πρόβλημα είναι ότι τα μεγάλα σκάφη ε, ανταγωνίζονται με μικρότερα Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Μακροπρόθεσμα. Θέλουμε λύση. Θέλουμε να βρούμε λύσεις που θα προσελκύσουν επενδύσεις. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Κύριε Βαντάλεν, καταλαβαίνω τι λέτε. Σε καλούς καιρούς δεν χρειάζονται τα αποθεματικά. Τώρα όμως κάτι πρέπει να κάνουμε. Σε περίοδο ισχνών αγελάδων δύσκολα τα πράγματα δεν υπάρχει πρόσβαση στα δάνεια και να σώσεις κάποιους που δεν τα πήγαν καλά ως επιχειρηματίες είναι δύσκολο τώρα γιατί δεν υπάρχει ρευστό. Έχουμε κάποια εμπειρία σε διάφορους φορείς, σε διάφορους οργανισμούς. Το πρόβλημα είναι το προσύνισμα του στόλου. Ένα από τα προβλήματα. Κάτι που θα επηρεάσει το στόλο των εσωτερικών, ε, της εσωτερικής Θέλουμε να κάνουμε οικονομίες Θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όμως μέσω βελτιώσεων. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των κινητήρων, να μπορούν να διαρκούν οι κινητήρες 10-15 χρόνια περισσότερο. Ίσως πρέπει να εξετάσουμε κινητήρες 500 ή 600 ύπων για να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό. Ίσως μπορούμε να μειώσουμε όμως και τον κυλινδρισμό των κινητήρων. Ίσως, γιατί ίσως δεν χρειαζόμαστε τόσο ισχυρού κινητήρες. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμμετάσχουμε στο πρασίνισμα του τομέα, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά το υγροποιημένο φυσικό αέριο δεν είναι συνταγή, δεν είναι η πανάκια, διότι η αποθήκευση αυτού του καυσίμου είναι κάτι δύσκολο. Και κυρίως τα μικρά σκάφη. Μία λύση είναι η μετασκευή σκαφών. Για να γίνει αυτό ε, όμως χρειάζονται πολλά χρήματα. Είναι πάρα πολύ δαπανηρή μετασκευή παίρνει ένα κινητήρα 5.000 ευρώ και πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλα τόσα για να μετασκευάσει τον κινητήρα. Κόστο εγκατάσταση κλπ. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμεί, σαν κλαδικό οργανισμό, είναι να αναπτύξουμε φθηνότερους μηχανισμούς μετασκευής. Ίσως αυτή είναι μια λύση. Όσον αφορά το άρθρο 8, το άρθρο 8 είναι αρκετά άκαμπτο όσον αφορά τους όρους που θέτει και προτείνω να συμπεριληφθεί εκεί πέρα και το πρασίνισμα. Να μία απάντηση που μπορώ να δώσω. Κάτι που θέλει η ESO είναι να υπάρχει καλύτερη συνεργασία. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, να εργαστούμε για το πρασίνισμα, χρειαζόμαστε όμως περισσότερη συνεργασία. Σε άσχημες εποχές δεν μπορούμε να βρούμε απαντήσεις για αυτά που συμβαίνουν στην αγορά καλές απαντήσεις. Μπορούμε όμως να αυξήσουμε τη συνεργασία. Αν το πετύχουμε αυτό, θα, ε, με ένα σπάρο θα πετύχουμε δύο τριγώνια, πιστεύω. Τώρα, η αποφυγή των συγκρούσεων πράγματι είναι ένα σημαντικό θέμα. Πρέπει Καμιά φορά από χώρα σε χώρα πρέπει να αλλάξει την πλευρά του ποταμού στην οποία πλέεις. Χρειάζεται λοιπόν σύστημα αυτόματο να μπορείς να, να βλέπεις που βρίσκονται τα πλοία. Χρειάζονται τεχνολογίες αποφυγής συγκρούσεων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θεολογάκη, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μας ξαναδίνετε το λόγο. Να τονίσω, θα ήθελα, κάποια σημεία λίγα σημεία από τα πολλά που αναφέρθηκαν και χαίρομαι πάρα πολύ διότι μας ε, δώσατε πάρα πολύ χρήσιμο υλικό. Καταρχάς ε, το θέμα της υποδομής. Φυσικά εξαρτώμαστε απόλυτα από τη νέα ε, δομή TNT και από το Connecting Europe για τα νέα έργα. Για συντήρηση χρειάζεται να υιοθετήσουμε μια άλλη στρατηγική και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική του Δούναβη και τη δουλειά που κάνει η Επιτροπή του Δούναβη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με αυτό. Και αυτό είναι μέρος του έργου που σκοπεύουμε να κάνουμε τις ερχόμενες ε, εβδομάδες και τους ερχόμενους μήνες. Να εντείνουμε δηλαδή τη συνεργασία έτσι ώστε όλα τα ε, ρηποαρικά κράτη να πληρούν τις ε, κατάλληλες προϋποθέσεις. Αναφέρθηκε επίσης ε, το ζήτημα της χρηματοδότησης. Φυσικά το, η διευκόλυνση στην στην Ευρώπη προβλέπει χρηματοδότηση για τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Μία, ένας τομέας είναι ε, εξοπλισμός τηλεματικής και από την άλλη πρέπει να δούμε τι γίνεται με ναι. τις βιώσιμες υπηρεσίες ε, μεταφοράς ε, φορτίου και πώς μπορούμε να εξυγχρονίσουμε τις μεταφορές αυτές. Τώρα όσον αφορά την καινοτομία δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ορίζοντα 2020. Επίσης τρέχει και το πρόγραμμα Πλατίνα, το οποίο έχει ένα περιεκτικότατο θεματολόγιο σχετικά με τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να απορροφήσουμε τη χρηματοδότηση. Τώρα όσον αφορά την ε, ένταξη σε έναν ενιαίο χώρο, να σας πω ότι το ΝΑΙΑΔΕΣ ε, είναι η πλατφόρμα όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η ένταξη και δεν είναι απλή σύπτωση. Εμείς έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ ε, στενά με όλους έτσι ώστε ε, να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Συνεργαστήκαμε με τη CCNR, με την Επιτροπή του Δούναβη που μας παρήχαν εμπειρογνωμοσύνη Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνεκτική ε, προσέγγιση για την εσωτερική ναυσιπλοεία η οποία βασίζεται στην ποιότητα η οποία με τη σειρά της ε, φαίνεται στο πρόγραμμα Ναϊάδα και στο έργο τη CCCR και τη Επιτροπή του Δούναβη. Εδώ φυσικά δεν θέλω να παραλείψω τι επιτροπέ του ΣΕΒΑ και του Μοζέλα οι οποίε επίση ήταν εξίσου σημαντικέ για την ε, ολοκλήρωση και την ένταξη του προγράμματος. Πρωτού ψηφίσετε, επιτρέψτε μου να πω κάτι τελευταίο, ότι όντως ε, υπήρξε δυσκολία στο να βρεθεί ομοφωνία. Αυτό που προσπαθούμε είναι να επεκτείνουμε, να διευρύνουμε τον κανονισμό έτσι ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες, ε, περισσότερες και γι' αυτό έχουμε συνεργαστεί και συνομιλήσει με όλους ε, τους ενδιαφερόμενους, με πάρα πολλούς τουλάχιστον έτσι ώστε να διασφαλιστεί αυτή η ομοφωνία, έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις για πρασίνισμα, να βρεθούν λύσεις για καινοτομία, λύσεις οι οποίες δεν θα παρεμβαίνουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν και αναμένουμε να υπάρξει ευρύτερη συμφωνία. Και αυτό θα οδηγήσει στην καλύτερη απορρόφηση αυτού του ταμείου, το οποίο αυτή τη στιγμή ύπταται και ορείται κάπου και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ε, μεγάλη στήριξη όλων ε, των μελών. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και επίση ε, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε στο ψήφισμά του να ε, αναφερθούν οποιαδήποτε άλλα ζητήματα θεωρεί αυτό χρήσιμα έτσι ώστε να έχουμε με ένα καλό μπούσουλο για το μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να σας πληροφορήσω ότι η κυρία Βόρτμαν Κόλ έχει δώσει προθεσμία για υποβολή τροπολογιών την 15η Ιανουαρίου. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή Μεταφορών στις 20 Φεβρουαρίου. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω τον Hans van der την Τερέζα Hacksteiner, τον Hank van der Welt, τους υπόλοιπους συνομιλητές για τη συνεισφορά τους στο δεύτερο πάνελ και να ευχαριστήσω ξανά και τους συμμετέχοντας στο πρώτο πάνελ. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας που ήρθατε παρακολουθήσατε την συζήτηση, συμμετείχατε και μας δώσατε την πυρογνωμοσύνη σας. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι στο μέλλον ελπίζω να δώσουμε ναι. μεγαλύτερη προτεραιότητα στις, ε, στην εσωτερική πλοία, διότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αναγκαίο για τις ευρωπαϊκές μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα σας. Ευχαριστώ λοιπόν όλους πάρα πολύ και θα συζητήσω τώρα κατεβείτε από το πόντιμ και εμείς θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας. Okay, can we go on with the next on the Να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έγγραφο εργασίας για την εσωτερήκευση και τη μείωση των και τη μείωση της εξωτερήκευσης του κόστου στις μεταφορές. Όλα αυτά συνδέονται με την ε, οδηγία περί ευρωβινιέτας ε, και το, η ομάδα των Πρασίνων ε, έθεσε το θέμα της συνέχειας στην οδηγία και θεωρεί ότι η της οδηγίας υπό το άρθρο 11.4 που λέει στις 16 Οκτωβρίου του 2012 η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει έκθεση που συνοψίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εσωτερήκευση ή τη μείωση του εξωτερικού κόστου σε σχέση με το περιβαλλοντικά και οικοθόρυβο και άλλες επιπτώσεις των μεταφορών. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει γιατί το δοκίμενο δημοσιεύθηκε με εννέα μήνες καθυστέρηση και υπό τη μορφή ενός εγγράφου, εσωτερικού εγγράφου εργασίας. Η απόφαση λοιπόν των συντονιστών στις 15 Σεπτεμβρίου ήταν να ζητήσουμε από την Κομισιόν να έρθει εδώ και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών της σε αυτό το τομέα. Ο κ. Σανταμάτο θα μας εξηγήσει λοιπόν που βρίσκεται η κατάσταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Η Κομισιόν έπρεπε να ανταποκριθεί στο αίτημα στην υποχρέωση τη οδηγίας ε, της για να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εσωτερική σε όλε τις μορφές μεταφορών. Ήταν μέγα ε, έργο. Ε, ζητήσαμε ε, από έναν όμιλο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων να μας βοηθήσουν, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέτρα τιμολόγησης για όλες ε, τους τρόπους μεταφορών. Μέτρα τιμολόγησης ε, που μπορούν να οριστούν πιο αυστηρά ως μέτρα εσωτερήκευσης. Το αποτέλεσμα είναι μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι, 700 σελίδες μελέτη. γίνεται λόγος εδώ για τους ε, δασμούς αλλά και την τιμολόγηση που χρησιμοποιούνται για την εσωτερήκευση των εξωτερικεύσεων. Επίσης, ένα αποτέλεσμα, βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία μέτρων για να μπορούμε να τα πάρουμε τα διάφορα μέτρα στους διάφορους τομείς ώστε να γίνει μια πραγματική εσωτερήκευση του ε, κόστους. Προκύπτει ότι περίπου το 2% του ΑΕΠ συλλέγεται ετησίως ε, κυρίως μέσω των δασμών επί των καυσίμων 1,4 του ΑΕΠ αλλά επίσης 0,5 μέσω της, ε, των, των φόρων κυκλοφορίας αυτοκινήτων αλλά και των ε, φόρων για τις πινακίδες. Ε, πολύ λίγα συλλέγονται από τα διόδια, 0,2 του ΑΕΠ μόνο. Η γενική εικόνα για τις οδικές μεταφορές είναι σχετικά ισορροπημένη Τώρα όσον αφορά την εξωτερήκευση για τις κλιματικές αλλαγές, αυτή καλύπτεται από τα φόρους στα καύσιμα, τους δασμούς μάλλον στα καύσιμα, ε, που αφορούν συγκεκριμένα σε εξωτερήκευση γιατί η εκπομπή ε, ρήπων από την κατανάλωση καυσίμων είναι εξωτερικευμένο κόστος, ενώ άλλα εξωτερικά κόστη όπως ε, μόλυνση του, των υδάτων ε, ή θόρυβος δεν λαμβάνονται υπόψη καταλήλως ε, οι δασμοί ε, καταγραφής ε, των οχημάτων δεν λαμβάνουν υπόψη το εξωτερικευμένο κόστος, δηλαδή δεν δίνουν κίνητρα, ενώ έχουμε βασικά την βινιέτα, αυτό το σήμα που βασίζεται σε χρονικά όρια, ε, όχι σε αποστάσεις. Θα ήταν αυτό ίσως πιο κατάλληλο να το αλλάξουμε. Η κατάσταση στις άλλες, ε, στα άλλα είδη μεταφορών είναι σχεδόν ανάποδη, αντίστροφη. Ε, δεν δίνεται έμφαση στις κλιματικές αλλαγές γιατί υπάρχουν μικρότεροι δασμοί στην ναυσιπλοΐα, αλλά και στην εσωτερική ναυσιπλοΐα Υπάρχει ε, συζήτηση για την ε, αεροπλοεία ενώ στους σιδηροδρόμους τα ηλεκτρικά τρένα ε, καλύπτονται μέσω του ETS αλλά αυτά τα τρένα έχουν εξαιρέσεις, χαίρουν μάλλον διαφόρων φορολογικών εξαιρέσεων. Τώρα, ε, στον, στους όλα τα κρατημέλη ε, χρεώνουν για τη φθορά των υποδομών και ορισμένα κρατημέλη για υψηλότερο ποσοστό κόστος των υποδομών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ε, οι δασμοί ε, χρήσης ε, σχετίζονται και με το θόρυβο, αλλά όχι σε αρκετό βαθμό ώστε να εσωτερικευθούν αυτά τα εξωτερικά κόστη. Στο θαλάσσιες μεταφορές παρατηρούμε τα αλμυνικά τέλη, τα οποία βασίζονται στο ΝΑΖ και στα φορτία. Κάποιες φορές τροποποιούνται και κυμαίνονται ανάλογα με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά των σκαφών. Ωστόσο, υπάρχει επίσης έλλειψη διαφάνειας για τις χρεώσεις για τα τέλη αυτά που κάποιες φορές ε, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις μεταφορικές εταιρείες και τις λιμανικές αρχές. Στην ε, αεροπλοεία τώρα έχουμε τέλη προσγείωσης και απογείωσης, τέλη που βασίζονται στους επιβάτες, κάποιες φορές ε, τροποποιούνται ανάλογα με το θόρυβο που παράγεται σε κάποιες ε, χώρες υπάρχει φόρος και στα εισιτήρια ε, αλλά δεν έχει προβλεφθεί και καμιά εσωτερήκευση. Τέλος, στις εσωτερικές πλωτές οδούς έχουμε λιμενικά τέλη παρόμοια με τα ε, θαλάσσια αλλά όχι στο Ρήνο και στο Δούναβι λόγω διεθνών συμφωνιών. Εν γέννη λοιπόν το μήνυμα που λαμβάνουμε από αυτή τη μελέτη ότι υπάρχει μάλλον ανεπαρκή σκάλυψη του εξωτερικού κόστους, αλλά υπάρχουν και πολλά έσοδα που συλλέγονται στις μεταφορές, αλλά τα οποία δεν συνδέονται με, με το εξωτερικό κόστος και άρα μια απλή εξισορρόπηση ή συλλογή των ίδιων εσόδων μέσω πιο διαφοροποιημένου συστήματος θα βελτίωνε γενικώ την κατάσταση. Αυτό είναι το τμήμα που αναφέρεται στους μηχανισμούς τιμολόγησης. Το αίτημα όμως της οδηγίας αφορούσε και ενημέρωση για τα ρυθμιστικά μέτρα. Τα αριθμιστικά μέτρα δεν είναι μέτρα εσωτερικευσής αυστηρά, αλλά βεβαίως έχουν αντίκτυπο για τα εξωτερικά κόστη, στα εξωτερικά κόστη, δεν δίνουν την επιλογή είτε να πληρώνονται είτε να ε, βοηθούν στις, στα εξωτερικά κόστη, ας πούμε βελτίωση ε, ε, προδιαγραφών ασφάλειας και για τα οχήματα κτλ. Και μάλιστα ένα μεγάλο τμήμα το κεκτημένο στις μεταφορές είναι επίπτωση μιας ε, κάποιου και από τα εξωτερικά κόστη. Το 2008 στο πλαίσιο του πρασινίσματος του πακέτου μεταφορών ε, ήδη εκπονήσαμε, να, κάναμε μια απογραφή μάλλον των ρυθμιστικών ε, μέτρων και τώρα μπορούμε να εστιάσουμε στα μέτρα που έχουν ληφθεί έκτοτε. Επίσης αναφέρομαι πτυχές που σχετίζονται με τις υποδομές και την έρευνα που είναι συμπληρωματικές σε μεγάλο βαθμό με τα μέτρα εσωτερήκευσης, δηλαδή η έρευνα για τις υποδομές δίνει εναλλακτικέ που καθιστούν το σήμα της ε, εξωτερήκευσης πολύ πιο αποτελεσματικό για την αλλαγή της νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Ελπίζω λοιπόν πως αυτή η μελέτη και η έκθεση θα σας δώσουν πολύ χρήσιμο υλικό για περαιτέρω σκέψη και προβληματισμό και αν θεωρείτε πως αυτά αρκούν ως εισαγωγή θα σταματήσω σε αυτά για την ώρα. Ευχαριστούμε κύριε Γκρός. Όχι, Ο κύριος Γκρός μάλλον θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση αυτή, για αυτό το έγγραφο εργασίας. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και για εμάς ε, φυσικά ε, είναι για πολλούς λόγους ε, γνωστό το περιεχόμενό της, όμως πιστεύω πως αυτό το έγγραφο βρίσκονται πάρα πολλά επιμέρους θέματα που είναι πολύ σημαντικό να επαναληφθούν και να αναλυθούν. Ε, έχουν γίνει ήδη πάρα πολλές συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό Σήμα Τελών Κυκλοφορίας ως ένα μέτρο αντιμετώπισης εσωτερήκευσης αυτών των εξωτερικών δαπανών, ως κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε μια ε, κοινή προσέγγιση. Αυτό όμως είναι αρκετά δύσκολο και γιατί, γιατί υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, διαφορετική φιλοσοφία στα κράτη-μέλη. Για πάρα πολλές ε, χώρες η εσωτερήκευση του, των εξωτερικών ταπανών ε, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την επικαιρότητα, το οποίο θα δώσει φυσικά επιπλέον έσοδα στα κρατικά ταμεία και θα μειώσει τις ταπάνες, όμως ε, συνδέεται άμεσα και με τις με άλλες ε, δομές και υποδομές, ε, για παράδειγμα κυκλοφοριακή συμφόρηση, περιβάλλον, δίκτυα μεταφορών. Έπειτα, δεν υπάρχει μόνο αντίθεση Ευρωπαϊκής Ένωση και κρατών μελών, αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωση και τρίτων χωρών. Εδώ σκέφτομαι για παράδειγμα την ε, θαλάσσια ναυσιπλοεία και τις αερομεταφορές. Ιδιαίτερα στι αερομεταφορές είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα ε, δράσουμε στο μέλλον, ποια προσέγγιση θα υιοθετήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε καταρχά πρώτα εδώ στο σπίτι μα και μετά προ τα έξω. Πιστεύω πως ε, είμαστε σε δυνατότητα να ε, δράσουμε συμβιβαστικά, όμως δεν θα μπορέσουμε SAE να δρούμε συμβιβαστικά. Επίσης, πιστεύω πως τα προβλήματα της εσωτερήκευσης του κόστους είναι κάτι που πρέπει να ε, δούμε ρεαλιστικά και όχι απλά ως ένα μέσο να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία. Επίσης πιστεύω ότι θα είναι προς το δικό μας ε, συμφέρον να συζητήσουμε το θέμα των αρμοδιοτήτων, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και να πω επίσης ότι στην έκθεση του Σαρίμελ Κατραουή αναφέρεται το περίφημο earmarking και το ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτή θα τους πραγματοποιήσει. Δεν πρέπει να είμαστε εδώ μόνο για να δημιουργούμε νέους φόρους που θα επιβαρύνουν τους πολίτες, αλλά και για να μπορούμε να τους βοηθούμε και να μειώνουμε επιπλέον έξοδα. Τώρα, διαβάζοντα την έκθεση, τι μπορώ να συμπεράνω. Μπορώ να συμπεράνω ότι έχουμε αρκετές δυνατότητες και χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι το έγγραφο αυτό θα μας απασχολήσει για τους επόμενους μήνε και θα μπορέσουμε, ελπίζω, να δώσουμε στους πολίτες κάτι χειροπιαστό και κάτι που θα βελτιώσει πολύ την εφισταμένη κατάσταση. Ο κύριος Ελκαντραούι. Ε, Ευχαριστώ, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά που μας είπε. Αλλά τελικά μείνανε κάποια κενά από αυτά που άκουσα. Είναι λυπηρό που για παράδειγμα δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τα προγράμματα κάποιων κρατών μελών. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια για την εσωτερική του εξωτερικού χρέους. Στο Βέλγιο να εφαρμόσουμε ένα σύστημα με εισφορές κατά χιλιόμετρο για τα φορτηγά. Κάποιες χώρες θα αναλάβουν παρόμοιες ε, πρωτοβουλίες. Θα είναι καλό να είμαστε ενήμεροι λοιπόν για το τι κάνει κάθε χώρα. Να ξέρουμε τι θα γίνει ε, στα πλαίσια της οδηγίας για αυτό το ευρωπαϊκό σήμα της Ευρωβινιέτας. Ε, αυτό είναι το πρώτο. Θέλουμε περισσότερες πληροφορίες πρώτα απ' όλα. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, έχουμε παρόλα αυτά κατά τρόπο μεταφοράς πληροφορίες όσον αφορά κάποιες πρωτοβουλίες, όσον αφορά τους φόρους, τις εισφορές που προβλέπονται, καλώς αυτό που θα ήθελα και αυτό που λείπει είναι πληροφορίες για την σχέση, τη θέση που έχει κάθε τρόπος μεταφοράς. Ποσοστά. Ποσοστά, αν καταλαβαίνετε θέλω να πω. γνωρίζουμε, και δεν νομίζω ότι γνωρίζουμε, γνωρίζουμε στα κράτη-μέλη τι προβλέπεται ε, για τους δρόμους, πράγματος χάρη. Ποιο κομμάτι του εξωτερικού κόστους καλύπτεται από τον καταναλωτή, από εκείνον που ρηπαίνει. Το ρωτάω αυτό, διότι αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες. Είναι κάτι που θα μπορούσε να ρίξει φως στη συζήτηση. για αυτού του είδου συζήτηση, το πρώτο ερώτημα είναι ότι αν τελικά υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Κάθε τομέας λέει ότι πληρώνει πολύ, το ξέρω. Πού βρισκόμαστε. Φόρος καυσίμων. Στοιχεία. Κατά μέσο όρο, από ό,τι μας λένε, 190 ευρώ ανατόνο ε, εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος. Ποιο είναι όμως το μερτικό κάθε ε, τρόπο μεταφοράς, πώς μοιράζεται αυτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί, αν είχαμε τα στοιχεία όμως θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στις ζητήσεις. Κάτι άλλο που λείπει. Και αφορά αυτό το τελευταίο κομμάτι του εγγράφου εργασίας. Θέλουμε πιο μεγάλη προσπάθεια από πλευράς ε, ε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Καλό αυτό. Όμως δεν έχουμε συγκεκριμένα κομβικά σημεία. Πού θα ευρισκόμαστε του χρόνου. Έχουμε μια λευκή βίβλο που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Στόχους για το 2020. Δεν θα είναι υποχρεωτική η εσωτερική του εξωτερικού κόστους. Θα είναι κάτι υποχρεωτικό. Αυτό είναι σαν στόχος του 2020. Τώρα δεν βλέπουμε όμως κάποια πράγματα. Κάποια άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να επαναλαμβάνονται και εδώ, αυτά που εμπεριέχονται στη Λευκή Βίβλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να προχωρήσει πιο πέρα, αυτό είναι το πρώτο μήνυμα. Μετά κάτι άλλο. Σε κάποια κάτι μέλη υπάρχει προβληματισμός όσον αφορά την αντιμετώπιση των ταχύ. Στη Γερμανία συζητείται αυτό, παντού λίγο πολύ. Έχω μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να κάνει ενδελεχή προβληματισμό επ' αυτού. Σήμερα τι λέμε στα κάτι μελη Λέμε, καλό θα ήταν να έχετε ένα σύστημα εισφορών ανά χιλιόμετρο, να εφαρμόζετε μέτρα στα πλαίσια της αρχής ο ρηπαίνων πληρώνει. Να αναλαμβάνει κάποιο κόστος ο καταναλωτής, εκείνος που ρηπαίνει, από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει αν ένα κάτω μέλος έχει τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να προβλέπει αποζημιώσεις, μειώνοντας το φόρο όσον αφορά το, τον φόρο για την αγορά ενός οχήματος. Και τα κράτη-μέλη έτσι στριμώχνονται. Άρα είναι ένα στοιχείο το οποίο αν είχαμε στοιχεία γι' αυτό θα μας βοηθούσε στη συζήτηση. Κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισνερ. Ε, οι δύο συνάδελφοί μου μίλησαν εκτενέστατα και αναφέρθηκαν και σε αυτά που ήθελα και εγώ να πω, οπότε θα είμαι σύντομη. Καταρχά, είναι πάρα πολύ καλό ότι έχουμε ένα έγγραφο, ότι έχουμε μια μελέτη. Από την άλλη, όπω είπε και ο κύριο Ακαντράου, έχουμε πάρα πολλά ε, πράγματα τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε. Πρέπει να ε, δούμε πω αυτό που στην ουσία μα λείπει είναι δασμευτικέ αποφάσει. Ε, είμαστε καλοί στα λόγια, αλλά όχι τόσο στι πράξει. όσον αφορά τη λευκή, η πράσινη βίβλο, ναι, φυσικά όλοι έχουμε του ίδιου στόχου για το περιβάλλον όλοι στη θεωρία είμαστε εντάξει. Το πρόβλημα είναι στην εφαρμογή αυτών των ε, στόχων και πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Γι' αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι μπορεί να κάνει, όχι μόνο να πει, αλλά να κάνει έτσι ώστε να φέρει τα κράτη-μέλη σε αυτή την ε, συμφωνία που θα οδηγήσει στην υλοποίηση των ε, στόχων. Από την άλλη, όσον αφορά το earmarking, την δέσμευση αυτών των κονδυλίων, Πώ μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συνένεση εδώ στο Κοινοβούλιο όσον αφορά το earmarking και στη, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο υπήρξε επίσης σε μεγάλη συμφωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά, ιδιαίτερα από τους ε, πολιτικούς ε, που ασχολούνταν με τις μεταφορές. Βλέπουμε όμως ότι δεν έχει εφαρμοστεί αυτό και ότι δεν έχουμε κοινή ε, οικονομική πολιτική. Και τι γίνεται με αυτό. Αυτό θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Λίχτεμπεργκερ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Συγγνώμη καταρχάς για την εργοπορία μου. Αυτό συμβαίνει συνέχεια με, όταν ε, πρέπει να είσαι σε πολλές ε, επιτροπές ταυτόχρονα. Κοίταξα όμως ε, τις παρουσιάσεις και την έκθεση και για μένα το ενδιαφέρον είναι το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε πραγματικά να κινήσουμε τα πράγματα και να τα κινήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα δύο ερωτήματα που καίνε και που είναι ακόμα άλυτα είναι η σχέσεις στο Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο υπάρχουν ορισμένες τάσεις. Να υπάρχει συμφωνία σε αρχικό στάδιο, μετά όμως να μη γίνεται τίποτα. Είχαμε και στη Γερμανία ε, και στην Αυστρία παρόμοιε ε, συζητήσεις. Ε, έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν επίση το, τα διόδια και εκεί υπήρχαν αρχικέ συμφωνίε στην πράξη όμως δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα, είναι σημαντικό καταρχάς να δούμε ότι πρέπει από τη μία ότι από τη μία μάλλον αποτρέπουμε τα κράτη-μέλη από το να ζητούν πολλά, από την άλλη όμως ζητούμε περισσότερη νομοθεσία. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Δεν μπορούμε να παρεμποδίζουμε συστηματικά την υλοποίηση αυτών που ζητούμε. Όλοι στα λόγια δεσμεύονται, στην πράξη όμως υστερούν. Αυτό λοιπόν ίσως σημαίνει ότι ζητάμε πολλά και αυτά είναι λίγα. Ίσως θα έπρεπε στο μέλλον να αλλάξουμε την στρατηγική αυτή. Θυμάστε και τις ε, ατέρμονες συζητήσει όσον αφορά την αεροπορία και το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Θυμάστε τι είχε γίνει και πόσο πολύ είχαν κρατήσει και τις ε, άλλες ε, συζητήσεις όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που εντείνονται με την χρήση της ενέργειας και πραγματικά να πω ότι έχω κουραστεί από αυτό το φαίνεστε. Τώρα, επί της ουσίας, θα ήθελα να ρωτήσω ποια βήματα προβλέπονται. Ξέρω πως είναι δύσκολο να απαντήθει κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε στο τέλος ε, θητείας, όμως ε, για μένα είναι σημαντικό να μάθω τι σχέδια υπάρχουν, πώς ε, σχεδιάζεται η υλοποίηση αυτών των σχεδίων ε, για, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα κράτη-μέλη. Ξέρω πώς ε, στα μέσα της χρονιάς θα αλλάξει η Επιτροπή, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι πραγματικά έχουμε στα χέρια μας και τι ανάγκες υπάρχουν και τι ανάγκες έχει το κάθε κράτος μέλος. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω για τις για τα σχέδια που υπάρχουν, εάν εσείς θεωρείτε πως μπορεί να συγκεντρωθεί μία πλειοψηφία, έτσι ώστε εάν δεν, κατα... δεν υπάρξει ομοφωνία τουλάχιστον να υπάρξει μία ίδια στάση, ίδια πολιτική επιθυμία. Είναι φυσικά κατανοητό και γνωστό ότι τα περισσότερα κράτη βρίσκονται σε μεγάλη οικονομική πίεση και πολλά από αυτά δεν καταφέρνουν να βρουν τα κονδύλια για να χρηματοδοτήσουν τον τομέα των μεταφορών. Από την άλλη όμως υπάρχουν απαιτήσει. Και αυτό πιστεύω ότι είναι από μόνο του μία αντίθεση Γι' αυτό λοιπόν να σας ενθυμίσω και την πρόταση που είχαμε κάνει στο παρελθόν να υπάρχει ανεξαρτησία από, την, ε, από τα διάφορα ταμεία, ιδιαίτερα στον τομέα της, ε, των μεταφορών ε, φορτίων μεγαλου βάρους. Έπειτα, τι θα γίνει με το περιβαλλοντικό κόστος, αμέ το κόστος ε, κάλυψης ε, ατυχημάτων. Αυτά θα με ενδιέφεραν να μάθω μεταξύ άλλων. Κύριε Ζουίκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω τα υποθέντα. Ερώτηση έχω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Που αφορά την προσημείωση ποσών. Μπορούμε να γνωρίζουμε, είναι δυνατόν, να γίνει μελέτη του θέματος για να γνωρίζουμε πόσα εισπράττει κάθε κάτος μέλος όσο για μέτρα υποδομών και εσωτερικεύσης του κόστους, πόσα εισπράττει από κάθε τρόπο μεταφοράς, πόσα χρήματα μέσω διαφόρων φόρων εισπράττονται από όλο το μεταφορικό σύστημα, αυτό από τη μία και από την άλλη πόσα ξαναδίνονται από αυτά τα κράτη για τις υποδομές και τα συστήματα βελτιώσεις ε, περιβαλλοντικής επίπτωσης των μεταφορών. Πραγματική ερώτηση. Είναι δυνατόν να υπάρχει ελάχιστη ε, ανάλυση αυτού. Ποια είναι η κατάσταση σε χώρες. 100% σε κάποιες χώρες από τους πόρους που εισπράττονται από τις μεταφορές δίνονται για βελτίωση των μεταφορικών υποδομών και για μέτρα για το περιβάλλον. Άλλες χώρες το 10% δεν ξέρουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό διότι μας ζητείτε να προβληματιστούμε και να προτείνουμε μέτρα σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσον αφορά τη φορολόγηση, τις προδιαγραφές, την υποστήριξη των υποδομών, ενώ η κατάσταση από χώρα σε χώρα, υποψιάζομαι, δεν ξέρω, πρέπει να είναι πάρα πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα. Και κλείνοντας θα πω ότι θα μπορούσαμε να δηλωτηθούμε μήπως θα πρέπει να έχουμε έναν δίκτυ. Ε, δίκτυ εισφορών που εισπράττονται και επιστροφή σε επενδύσει από χώρα σε χώρα. Είναι αδύνατο να ζητείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεσπίζουν ε, μέτρα σε τέτοια κλίμακα όταν δεν γνωρίζουν καθόλου τα θεσμικά όργανα ποια είναι η χρήση αυτών των χρημάτων. Και πιστεύω ότι διαφέρει πάρα πολύ κατάσταση από χώρα σε χώρα. Όσον αφορά τι υποδομέ, υπάρχει ευρωπαϊκή διάστοση και προστιθέμενη αξία όσον αφορά τι υποδομέ. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό, θα το επαναλάβω. Όσον αφορά τη ρήπανση εκπομπέ, αυτά δεν σταματούν στα σύνορα και θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ακαταστασία όσον αφορά την ίσπραξη τελών και μετά τον προορισμό των χρημάτων που εισπράττονται. Κύριε Σαντομάτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις, ξεκινώντας από το τελευταίο σημείο, το earmarking, την προσημείωση των ποσών. Στη μελέτη αναφέρεται ποιες μορφές ίσπαξης τελών ή ε, φόρων ε, σε διάφορα κάτι μέλη. Δεν υπάρχουν παραδείγματα πολλά. Ο φόρος στις ασφαλίσεις που έρχεται στο μυαλό που πολύ συχνά αυτά τα χρήματα πηγαίνουν ε, σε θέματα ασφαλείας των ε, χρηστών. Το θέμα αυτό του earmarking, ε, η προσημείωση των πόρων είναι κάτι και πώς γίνεται η κατανομή των πόρων δεν καλύπτεται πολύ καλά. Εμεί ζητούμε να γίνει κάτι τέτοιο μέσω της οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα, αλλά υπάρχουν στεναρές αντιδράσεις από κάποια κράτη-μέλη. Κάτι άλλο δυσκολότατη συλλογή στοιχείων, κυρίως εκτός του δικού τομέα. Η μελέτη προήλθε από έρευνα. Ερευνήσαμε την κατάσταση σε μεγάλα αεροδρόμια, σε μεγάλα λιμάνια, αλλά είναι σχεδόν αδύνατον να συλλέξουμε στοιχεία για όλες τις υποδομές τις μεταφορικές και όλα τα τέλη που επιβάλλονται στον τομέα αυτό σε τοπικό επίπεδο, οι γέφυρες, σύραγγες, ε, ε, φράγματα σε εσωτερικά συστήματα ναυσιπλοείας. Εκεί σπράττω διάφορα τέλη. Πολύ δύσκολο λοιπόν να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τον τομέα. Εξίσου δύσκολο είναι να κάνουμε πλήρη σύγκριση της καταστάσεως που επικρατεί στους διάφορους ε, τρόπους μεταφορών και να πούμε ποιος πληρώνει περισσότερα για εξωτερήκευση κλπ. Επίσης διότι η κατάσταση διαφέρει πολύ από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που απορρέει από την μελέτη. Ξέρω ότι αυτή δεν είναι η απάντηση που θέλει να λάβει κανείς. Θα θέλαμε κι εμείς να έχουμε καλύτερη ε, συγκρισιμότητα των στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τρόπους μεταφορών. Αλλά προσεγγίζοντας το πρόβλημα με τρόπο τέτοιο που να έχει στόχο την, ε, τον ιδεώδη, τον ιδανικό ανταγωνισμό ε, είναι κάτι δύσκολο. Υπάρχουν, ε, βλέπετε, τόσα πολλά στοιχεία πρέπει να λάβουμε υπόψη και, διαφοροποίηση ενός, και υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ τομέων. Καλύτερα να προχωρήσουμε προς συμπερίληψη περισσότερων Μεγαλύτερη συμπερίληψης της ένεσης εσωτερήκευσης στις διάφορες πρωτοβουλίες και στους διάφορους τρόπους είναι κάτι πιο εύκολο. Βήμα-βήμα να προχωράμε. Με αύξηση της εσωτερήκευσης και πράγματι αυτό θέλει να κάνει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο για μένα να πω οτιδήποτε που ξεπερνά το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το αναφέρουμε στη μελέτη. Πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο, δεν άλλαξαν οι στόχοι. Η Λευκή Βίβλος επανέλαβε τα υποθέντα στο πακέτο πρασινίσματος των μεταφορών του 2008. Η πολιτική εξακολουθεί να είναι πολιτική που έχει σαν ύψιστη προτεραιότητα, μία από τις μεγάλες προτεραιότητες στην εσωτερήκευση του κόστους. Αυτό είναι σημαντικό για πολλές πτυχές και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να προωθήσουμε αυτή την αρχή σε περαιτέρω πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε κλείνουμε και αυτό το θέμα. Να υπενθυμίσω στα μέλη ότι χώρος και το, ο τόπος και χρόνος Επόμενη συνεδρίαση είναι 20 Ιανουαρίου, 5η, 3 η ώρα. Δευτέρα, νομίζω ότι είναι. Δευτέρα 20. Δευτέρα, Δευτέρα. Όχι Πέμπτη, Δευτέρα. Δευτέρα λοιπόν. 20 Ιανουαρίου. Εύα. Σύντομη παρατήρηση. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιορίστηκε σε μόνο λίγα σημεία και παρέλειψε πάρα πολλά τα οποία θα θέλαμε να μάθουμε, τα οποία είχαμε ζητήσει να μάθουμε, το πώς θα συνεχίσουμε δηλαδή και λοιπά. Και αυτό δεν ήταν ερώτηση μόνο δική μου, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί και να μας απαντήσει γραπτός. Δίκιο αίτημα, αν μπορούσε να το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μου στείλει γραπτός απαντήσεις και να τις διαβιβάσω στους συντονιστές. Σαΐντ. Yes, uh, you, Ευχαριστώ για την ευελιξία σας, Πρόεδρε. Κάτι άλλο, παρατήρηση. Σε αυτό το θέμα, αλλά και σε άλλα πολλά, το θέμα των στοιχείων είναι σημαντικό. Όταν μιλάμε δικαιώματα επιβατών, για τέτοια θέματα. Προτείνω στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λαμβάνει αυτό υπόψη στις νομοθετικές της προτάσεις. Η συλλογή στοιχείων και η αναρμόνιση αυτής πρέπει να είναι θέμα. Είναι σημαντικό. για να μπορούμε να συζητούμε με σωστό τρόπο και στο μέλλον. Να λαμβάνετε υπόψη. Κύριε Σανταμάτο, θέλετε να απαντήσετε. Το θέμα των στοιχείων, συλλογής των στοιχείων, βεβαίως, τι να πω, υπάρχει μεγάλη, μεγάλη ανάγκη στοιχείων για να θεσπίσουμε νομοθεσία σωστή και φυή. Απ' την άλλη θέλουμε να μειώνουμε το διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις. Άρα αυτό δημιουργεί εντάσεις από τις δύο πλευρές. Διότι ο τομέας θέλει να μειώνονται οι απαιτήσει νομοθετικές για την παροχή στοιχείων. Συμφωνούμε απόλυτα. Θα θέλαμε περισσότερα στοιχεία. Αλλά, αλλά υπάρχει αυτή η ένταση μεταξύ των δύο αναγκών, των δύο πλευρών. Το επόμενο βήμα. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται νέα πρόταση για τα οδικά τέλη, τέλη κυκλοφορίας, που θα αντικαταστήσουν αυτά τα ειδικά σήματα ε, που επιβάλλουν τέλη με βάση τις αποστάσεις και για τα γιοταχή. Υπάρχει μια πρωτοβουλία για το θόρυβο που παράγεται από τη μεταφορά φορτίων σιδηροδρομικός. Θέλουμε να θεωρήσουμε την οδηγία για τα κινούμενα μηχανήματα εκτός δρόμων ε, κάτι που αφορά ίσως και τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοείας και με την ΙΚΑΟ εξετάζουμε και το θέμα του ETS για τα αεροσκάφη συστήματα για τα αεροσκάφη και το σύστημα ελέγχου, επαλήθευσης και ενημέρωσης και κοινοποίησης για τις εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές. Επ' αυτόν ε, κινούμεθα. Φοβάμαι ότι, ότι δεν μπορώ να πω περισσότερα. σχετικά με αυτό που έχουμε μπροστά μας και κουβεντιάζουμε. Ευχαριστώ. Καλώς λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, 20 Ιανουαρίου στις 3 το απόγευμα η επόμενη συνεδρίαση. Πάμε στους συντονιστές και όσοι δεν πρέπει να είναι παρόντες σα αποχωρήσουν. Θα είναι γρήγορη συνεδρία, σύντομη των συντονιστών. Παρακαλώ όσοι είναι να αποχωρήσουν να σας αποχωρήσουν.